Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα βασιστούμε στους διερμηνείς για να βγάλουν νόημα από αυτά που θα λέω. Σημαντικότητα εκκράση. Ο Μάικλ Κάσμαν είμαι εγώ. Είμαι αρχικό ε, εισηγητή για τον κανονισμό για την πρόσβαση του κοινού στα κοινά, κανονισμό 1049 του 2001 και είμαι εισηγητή του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αθέωση του κειμένου. Θα είμαι συντομότατο διότι το πρωινό εγχείρημα είναι να ακούσουμε τους φιλοξενούμενους, τους επισκέπτες, ε, να ακούσουμε τι έχουν να πούν όσον αφορά την αναθεώρηση και το πόσο σημαντικός είναι ο κανονισμός 1049. Να θέσω το πλαίσιο την ακρόαση. Θα το θέσω το θέμα στον Κρας τον το Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Θα σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ότι έγινε μια προσπάθεια να σταματήσουν αυτή την ακρόαση σήμερα το πρωί. Ποια ήταν η δικαιολογία ότι δεν συμμορφωθήκαμε στο τελικό κανονισμό όσον αφορά την κοινοποίηση των συνεδριάσεων και το θέμα τέθη στην ημερήσια διάταξη του Προεδρείου προς απόφαση ανευσυζητήσεως. Αυτό καθεαυτό νομίζω ότι δείχνει ανησυχητική τάση στο ύψιστο επίπεδο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τη δυνατότητα που θα μπορεί να έχει το κοινό να ελέγχει τα θεσμικά όργανα. Θα σταματήσω εδώ, δεν θα δημιουργήσω θέμα. Θα δώσω το λόγο σε συνάδελφο συγκητή της Συνταγματικής Επιτροπής. την Ανελή Γιατεμονακή. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πολύ χαρούμενη που διοργανώνω αυτό το σεμινάριο με καλούς ε, συναδέλφους, τον Μάικλ Κάσμαν και την κυρία Χαουτάλα Όλοι μας εργαστήκαμε για μια διαφανέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση επί μακρόν. Στις προσπάθειές μας καμιά φορά πετύχαμε, καμιά φορά, κάποιες φορές αποτύχαμε, αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε. Όλοι στην αίθουσα γνωρίζουν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Όμως, καταρχάς, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαφάνεια, γιατί είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα, διότι καμιά φορά λησμονούμε το βασικό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε να εφαρμόζεται η δημοκρατία, να ισχύει η δημοκρατία. Διότι αν δεν γνωρίζει κανείς πολλά, αν δεν μπορεί να συζητήσει, δεν μπορεί, δεν να χρησιμοποιήσει τα δημοκρατικά μας εργαλεία. Παραδείγματος χάρη για την ψηφοφορία, για να ψηφίσει. Δεύτερον, θέλουμε να προωθήσουμε την ορθή διακυβέρνηση. αυτή είναι οι δύο βασικοί στόχοι. Και με θλίψη μου λέω ότι η οδηγία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απομακρύνει τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέλουμε αυτό. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες περί του τι δεν γενέστε. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πρόταση οδηγίας, όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε κοινοτροπίες τον τρόπο του σκέπτεστε. Δεν αρκεί να κατατεθεί η οδηγία, η νοοτροπία είναι το σημαντικότερο να αλλάξει. Είναι και το δυσκολότερο όμως. Χρειάζεται χρόνο. Και καμιά φορά δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Όμως, αν θέλουμε δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε επίσης πραγματική διαφάνεια πάνε χέρι με χέρι. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στη δέσμευση που ανέλαβε για τη διαφάνεια. Πρέπει να προωθήσουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την ορθή διακυβέρνηση. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη. Χαίρομαι που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις παρούσες, διότι ξέρω ότι για να αυξηθεί η διαφάνεια, η ανοιχτή προσέγγιση και η πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χρειαζόμαστε όλος ιδιαίτερο την υποστήριξη των μη κυβερνητικών φορέων, της οργανώσεις δημοσιογράφων, τους ιδιώτες ε, δημοσιογράφους. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, να βρούμε νέους τρόπους για να προχωρήσουμε. Είστε ευπρόσδεκτοι, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ανελή. Χάιντι Χάουταλα να κάνει κάποια πρώτα σχόλια και μετά να προεδρεύσει του πρώτου τμήματος συνεδριάσεως. Λοιπόν, Χάιντι, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, όπως είπε και η Ανελή. Η συνεισφορά και η πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανοιχτή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σημαντικότατη. Πάντα ήταν σημαντική. Θυμούμε όταν κάποιοι από εμά διοργανώσαμε μία κρόαση εδώ στο Κοινοβούλιο την άνοιξη του 1999 ανακαλύψαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διοίκηση ευρωπαϊκή δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουν το, και ότι πρέπει να έχουν το πλήρως δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτό υπογραμμίστηκε από μία φράση που ανακαλύψαμε σε μία ανεπίσημη ανακοίνωση μαζί με τον Τόνι Μπάνι και άλλους που έλεγε ευθέως ότι θα ήταν αναγκαίο να αποφευθεί η περίπτωση κατά την οποία οι πολίτες θα μπορούν να παρεμβαίνουν στις λήψεις αποφάσεων. Αυτό για μένα με την πάω των ετών αντιχούσε στο κεφάλι μου. Όποτε σκέφτομαι επόμενα βήματα αυτό σκέφτομαι και οι τρεις μας είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που σας βλέπουμε εδώ στην αίθουσα παρόντες διότι πρέπει να ξεπεράσουμε την αποτελμάτωση της τελευταίας διετίας όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουμε και είμαι πολύ χαρούμενοι που δίνω που έχω την πρώτη δυνατότητα να εξηγήσω πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα. Και χαίρομαι που ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος είναι εδώ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, που έχει πετύχει πάρα πολλά στον τομέα αυτό της συμμετοχής των πολιτών στην ε, λήψη αποφάσεων και συνεπώς το δικαίωμα να γνωρίζουν τα τεκτενόμενα. Κύριε Διαμαντούρο, παρακαλώ να πάρετε το λόγο και σας προειδοποιώ όλους ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί εμείς οι πρόεδροι όσον αφορά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Ε, δεν θα υπάρξει ίκτος για κανέναν. Θα είμαστε άτεγκτοι. Έχετε το λόγο κύριε Διαμαντούρο. Ευχαριστώ πρόεδρε λαμβάνω υπόψη το γεγονό θέλετε να είσαστε άπονοι. Δεν σας γνωρίζω ως άπονοι, αλλά θα το δεχτώ. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν μπω στις παρατηρήσεις μου, θα ήθελα ε, με δυο λόγια να πω ότι ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, αλλά και ως πολίτης, συμφωνώ 100% με τις ε, παρατηρήσεις Τη κυρίας Χάουταλα και της κυρίας Μάκη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάγκη αλλαγή νοοτροπία. Αυτό αποτελεί όρο και συνθήκη προκειμένου οι πολίτες να χαίρουν πλήρους πρόσβασης. Ε, και ε, να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και της, ε, την κυρία αλλά την κυρία Γιάτενμά και τον κύριο Κάσμαν που οργάνωσαν αυτή την ακρόαση. Η ακρόαση αυτή έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ και καιρό. Μου ζήτησαν να μιλήσω για το τι έχουμε μάθει από τις προσφυγές των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι έχουμε μάθει, μπορούμε να μάθουμε πέντε κυρίως πράγματα. Πρώτον, είναι ότι λίγοι πολίτες γνωρίζουν ότι η συνθήκη της Αβώνας διευρύνει το δικαίωμα της ε, ε, πρόσβασης σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, υπηρεσίες και ε, θεσμικά όργανα. Ορισμένοι, μάλιστα, ορισμένα μάλιστα από αυτά τα όργανα και τις υπηρεσίες αγνοούν και, και τα ίδια το γεγονός. Από εδώ και πέρα θα μιλάω για θεσμικά όργανα μόνον και θα τα περιλαμβάνω όλα αυτά και τα γραφεία και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Οπότε θα... Ε, Είμαι και πιο γρήγορο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Προτείνω να ξεχωρίσουμε αυτό το πρόβλημα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, ε, τα οποία προκύπτουν από τη συζήτηση για την ε, πρόταση τη Κομισιόν που έγινε πριν από τρία χρόνια για την ε, αναθεώρηση του κανονισμού, για την αδιατύπωση του κανονισμού 1049-2001. Στο Κολέγιο των Επιτρόπων, στι 15 Φεβρουαρίου, όταν είχα προσκληθεί εκεί, είχα προτείνει στην Κομισιόν να υποβάλει μια περιορισμένη πρόταση αναδιατύπωση του κανονισμού κανονισμού για να ληφθεί απλώ υπόψη η συνθήκη τη Λισαβόνα. Χαίρομαι που η Κομισιόν έχει υποβάλει πλέον μια τέτοιου είδου πρόταση. Ελπίζω ότι αυτέ οι μικρέ περιορισμένε αλλαγέ, οι οποίε δεν δημιουργούν ε, αντιθέσει και προβλήματα, ε, θα μπορούσε να, ρυθμίσει, να, θα μπορούσε να υιοθετηθεί γρήγορα. Ε, δεύτερον, σε όλες τις προσφυγές ε, τις οποίες έχω εξετάσει δεν βρήκα ούτε μία περίπτωση στην οποία να πιστώ ότι οι εξαιρέσει στο δικαίωμα πρόσβασης είναι τόσο πολύ στενές που δεν επιτρέπουν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρεται αυτό στο άρθρο 4 του κανονισμού. Αντιθέτως μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις που, στις περιπτώσεις που εγώ ε, εξέτασα και που ε, θεωρήθηκε ότι το, η χορήγηση του δικαιώματο πρόσβαση θα ε, δημιουργούσε, προκαλούσε βλάβη, ε, δεν, μία τουλάχιστον από τι εξαιρέσει πάντοτε εφαρμοζόταν. Οπότε δεν υπάρχει θέμα διεύρυνση των εξαιρέσεων. Το τρίτο σημείο, που, το τρίτο δίδαγμα αφορά το θέμα των καθυστερήσεων της Κομισιόν να χειριστεί ε, τις αιτήσει. Πολύ συχνά η Κομισιόν λέει ότι καθυστερεί επειδή το κάποιο κράτος μέλος δεν απάντησε έγκαιρα όταν του ζητήθηκε η γνώμη του για την πρόσβαση σε ένα έγγραφο το οποίο προκύπτει, προέρχεται από το ίδιο το κράτος μέλος. Σύμφωνα με την ομολογία θα πρέπει να ε, λαμβάνει η χώρα ένα γνήσιο διάλογο ανάμεσα στην Κομισιόν και το κράτο μέλο. Όμω δεν πιστεύω ότι ο γνήσιο διάλογο θα πρέπει να οδηγεί ε, σε μακρέ καθυστερήσει εις βάρος του θεμελιών δικαιωμάτων των ε, πολιτών για την ε, πρόσβαση, όπως αυτό καθορίζεται από τη Συνθήκη και το, τη Χάρτα των θεμελιών Δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι η Κομισιόν ε, θα συμφωνήσει ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί όμοιρο των διαβουλεύσεων αυτών με το κράτο μέλος. Το τέταρτο δίδαγμα είναι το εξή, ότι τα θεσμικά όργανα δεν έχουν λύσει ακόμα το πρόβλημα του προσωπικού ε, που χρειάζεται για να ε, εξασφαλιστεί το δικαίωμα αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1049, αν μια αρχική αίτηση απορριφθεί εν μέρει εν όλο ή ελήψη απάντησης από το θεσμικό από το όργανο μπορεί να κατατεθεί επιβεβαιωτική αίτηση. Αν και αυτή απορριφθεί ε, μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο ή στον ε, διαμεσολαβητή. Ένα από τα κλειδιά για την καλή διαχείριση συστήματος είναι η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων που ε, τα έγγραφα ε, απελευθερώνονται μόνο μετά την επιβεβαιωτική αίτηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκε... υπάρχει αρκετό εκπαιδευμένο προσωπικό ε, για να απαντάει γρήγορα και με ακρίβεια στι αιτήσει. Το άλλο κλειδί για την καλή διοίκηση είναι να αποφύγουμε την ανάγκη ακόμα και για αρχικέ αιτήσει. Αυτό πώ μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει όταν εκ των προτέρων μπουν, ε, δημοσιεύονται ε, τα έγγραφα και οι πληροφορίε που χρειάζονται οι πολίτε. Μία από τι προτάσει που έκανα για την η βελτίωση διαχείρισης του δικαιώματος της ε, ελεύθερης πρόσβασης είναι ότι κάθε όργανο θα πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον άτομο ε, υπεύθυνο για την, ε, την χορήγηση πληροφοριών θα έχει το δικαίωμα διαχείριση αυτού του και θα έχει την ευθύνη διαχείριση αυτού του δικαιώματο θα φροντίζει να ε, απαντάει γρήγορα στις αιτήσει, να δικαιολογεί τις αρνήσεις και εκ των προτέρων να θέτει τα παρέτα έγγραφα ε, σε δημόσιο χώρο. Ε, επίσης θα μπορούσε να έχει ένα εκπαιδευτικό ρόλο που θα εξηγεί τους νομικούς κανόνες κλπ και τα ωφέλη από το να λειτουργούμε ανοιχτά. σας ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας ε, ε, Δεδομένων δημοσίευσε στις 24 Μαρτίου ένα κατευθυντής γραμμές για τις σχέσεις ανάμεσα στην ελεύθερη πρόσβαση και την προστασία των δεδομένων θα, ενώ υπό το της απόφασης της, της Bavarian Lager το, η υπηρεσία αυτή ζητάει από τα ε, θεσμικά όργανα να έχουν μια τέτοιου είδους ε, προορατική προσέγγιση. Ε, η υπηρεσία αυτή λέει ότι υπάρχουν περίπλοκες καταστάσεις όπως η περίπτωση Bavarian Lager που ε, τα θεσμικά, τα όργανα ε, περιμένουν μια αίτηση για, πρόσβαση πριν ε, σκεφτούν τι θα κάνουν με τις πληροφορίες που διαθέτουν. Θα πρέπει να είμαστε προορατικοί λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση αυτή του EDPS, του Επόπτη Προστασίας και μάλιστα πιστεύω ότι η καλή διοίκηση απαιτεί από τα όργανα να είναι προορατικά όχι μόνο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αλλά και σχετικά με άλλα συμφερόντα που προστατεύονται από το άρθρο 4 του 1049 και αυτό είναι το πέμπτο δίδαγμα. Πιο συγκεκριμένα, έχω πιστεί ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι προορατική και να διασφαλίζει ότι ε, τρίτα μέρη, συμπληρωμένων και των κρατών μελών, καταλαβαίνουν ότι ο βασικός κανόνας είναι η ελεύθερη πρόσβαση. Ένα τρίτο μέρος που δίνει ένα έγγραφο στην Κομισιόν θα πρέπει να εντοπίζει οποιοδήποτε τμήμα του για το οποίο, αφορούν, ε, ε, για το οποίο ισχύουν εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 και να το δικαιολογεί. Ταυτόχρονα με την αποστολή του εγγράφου στην Κομισιόν, από την Κομισιόν από την μεριά της θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά όταν λαμβάνει έγγραφα ότι αυτές οι απαιτήσει έχουν τύχη συμμόρφωσης. Αν όχι θα πρέπει αμέσως να λαμβάνει δράση έτσι ώστε να γίνουν σεβαστοί. Ε, αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό ότι οι πολίτες οι οποίοι ζητούν πρόσβαση έχουν, βλέπουν τα δικαιώματα προστατεύονται και ταυτόχρονα θα προστατεύεται και το δικαίωμα στην καλή διοίκηση. Ε, είμαι πεπισμένο ότι θα ήταν χρήσιμο ο κανονισμό 1049 να τροποποιηθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και προθεσμία για τα κράτη-μέλη να απαντούν ε, στι διαβουλεύσει και πιο ισχυρέ απαιτήσει ε, προορατικότητα. Παρ' όλα αυτά, κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποια καινούργια νομοθεσία. Τα όργανα και ιδιαίτερα οι Κομισιόν θα μπορούσαν ήδη να ξεκινήσουν δράση τώρα για να εφαρμόσουν το θεμελιώδη δικαίωμα της ελεύθερης ε, πρόσβαση πιο αποτελεσματικά. Ε, θα μπορούσαν ε, να ορίσουν information officers με καθήκον όπως αυτό που, αυτό που είπα προηγουμένω δηλαδή να απαντούν γρήγορα και με ακρίβεια και να προωθούν μια προορατική προσέγγιση στη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντούρα. Όλοι σημειώνουμε λοιπόν ότι δεν ε, χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι να φτάσει η νέα νομοθεσία. Και περνάω τώρα στην Αναή που εκπροσωπεί την Client Earth, που είναι μία από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της και που έχουν αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα όταν προσπαθούν ε, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για να ακούσουμε τι σημαίνει πρόσβαση στα δεδομένα όταν οι πολίτες αρχίζουν να χρειάζονται τα δεδομένα και ζητούν πρόσβαση στα έγγραφα. Αναής Μπερτιέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτή την ακρόαση και που μας προσκαλέσατε για να μιλήσουμε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όταν εμεί υποβάλλουμε αίτημα για να έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δύο λόγια να σα πω ότι η Client Earth είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από νομικού και χρησιμοποιούμε τον τομέα του δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, είναι σημαντική για μας η, προστασία, η πρόσβαση στα δεδομένα και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια γενικευμένη συμπεριφορά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μην δίδουν τα έγγραφα τα οποία θα έπρεπε να είναι προσβάσιμα χωρίς να δίνουν και κάποιου, κάποιες ισχύουσες δικαιολογίες ε, και αυτό πρόκειται για θεματικά έγγραφα ή για γενικότερα έγγραφα. παραβιάζεται η σύμβαση του Όρχους και δεν τηρείται η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας περιγράψω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο κανονισμός 1049 δεν είναι συμβατός με τη Σύμβαση του όρχου. Η Σύμβαση του όρχου είναι μια διεθνής σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες και για την συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση τη δικαιοσύνη σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του όρχου το 1985 και επομένως είναι δεσμευτική η Σύμβαση του Όρχου για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωση Επομένως, η σύμβαση του Όλχους ε, υπερισχύει ε, έναντι ε, άλλων ε, νομικών κειμένων και υπερισχύει του κανονισμού για την πρόσβαση σε δεδομένα. Υπάρχουν εξαιρέσει βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού που δεν επιτρέπονται βάσει τη Σύμβαση του Όρχου. Παραδείγματο χάρη, η Σύμβαση του Όρχου δεν επιμένει την παρακράτηση δεδομένων σχετικά με την οικονομική πολιτική μια χώρα, δεν επιτρέπει την μη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με νομικέ συμβουλέ ή έρευνε σε ποινικά ή πειθαρχικά θέματα. Εκτός από ποινικά ή πειθαρχικά θέματα. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δεν δίδουν πληροφορίες βάσει των εξαιρέσεων του άρθρου 4, αλλά βάσει της σύμβασης του όρχους αυτό είναι παράνομο. Όμω όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί στου οποίους υποβάλλουμε αιτήματα για να έχουμε πληροφορίες βασίζουν την άρνησή τους σε αυτές τις εξαιρέσει του άρθρου 4. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι παράνομες. Ε, Ω αποτέλεσμα πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε τρει υποθέσει τώρα ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη επιτροπή και μία υπόθεση κατά του Συμβουλίου. Αυτή η αναδιατύπωση του κανονισμού αποτελεί λοιπόν ευκαιρία για να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τη σύμβαση του Όρχους. Γιατί είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχίζεται, να έχουμε ένα παράτυπο κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να είναι συμβατή με τη σύμβαση του Όρχους. Πριν πριν από ένα μήνα η Επιτροπή Ελέγχου Συμβατότητας τη Σύμβασης του όρχου, διαπίστωσε ότι, δεν, ότι αν δεν αλλάξουν οι διατάξεις αυτές, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι συμβατή με τις διατάξεις της Σύμβασης του όρχου σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό πρόβλημα συμβατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σύμβαση του όρχου και η αναδιατύπωση του κανονισμού είναι ευκαιρία να προσαρμοστεί η συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σύμβαση του Όρχους. Δεύτερον τώρα, στις περισσότερες απαντήσεις που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι δεν, είναι, δεν συμμορφούνται με τον ε, κανονισμό και βασικά με τι χρονικές προθεσμίε που αναφέρονται στον κανονισμό. Η Επιτροπή ζητά συστηματικά χρονικές παρατάσει, ακόμη και αν δεν υπάρχει τίποτα που να αιτιολογεί τη χρονική παράταση. Ακόμη και αν ένα αίτημα δικό μας δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή ιδιαίτερα ογκώδες. Μερικές φορές έχουμε το πρόβλημα ότι δεν απαντούν καν στις επιβεβαιωτικές μας αιτήσει. Ε, ως εκ τούτου, δεν έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία ζητάμε εγκαίρως και αυτό μας εμποδίζει να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να έχουμε πραγματική συμμετοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Δεν μας επιτρέπει καν να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν, να καταλάβουμε τα θέματα περί των οποίων ε, πρόκειται και να μπορούμε να συμμετάσχουμε ενεργά. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και όπως είπε και ο Διαμεσολαβητής, ε, η Επιτροπή και ε, τα θεσμικά όργανα δεν δίνουν τις πληροφορίες οι οποίες θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες είναι πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες. Παραδείγματος χάρη μελέτες για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη κάποιες περιβαλλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστημονικές μελέτες, παραδείγματος χάρη για την επίπτωση των βιοκαυσίμων στην κλιματική αλλαγή. Αυτές είναι πληροφορίες που θα έπρεπε να διαχέονται από την Επιτροπή με ενεργό τρόπο όχι μόνο να είναι διαθέσιμες κατόπιν ετήσεω. και αυτές οι πληροφορίε δεν είναι καν διαθέσιμες κατόπιν ετήσεω. και αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να βελτιωθεί. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι πολλές από τις απαντήσεις που λαμβάνουμε δεν συμμορφούνται με την ομολογία του δικαστηρίου. Ακόμη λοιπόν και όταν υπάρχουν αποφάσει που έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επί των οποίων θα μπορούσε να βασιστεί η κοινωνία των πολιτών καθώς και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα είναι αποφάσεις με τι οποίες δεν συμμορφούνται τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένω πρέπει να καταφύγουμε και πάλι στο δικαστήριο για να επανεπιβεβαιώσει το ίδιο το δικαστήριο τι δικέ του αποφάσει. Παραδείγματο χάρη σε μια υπόθεση που κρεμεί ενώ, ε, ενώπιον του δικαστηρίου κατά του Συμβουλίου έχουμε ζητήσει να έχουμε πρόσβαση στη νομική γνωμοδότηση τη νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου για το παραδεκτό της τροπολογίας του Κοινοβουλίου για την πρόταση τη Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση αυτή που συζητάμε. Δηλαδή ε, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με την υπόθεση Τούρκο. Σχετικά με νομοθεσία που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη προς το κοινό. Το Συμβούλιο αγνοεί εντελώς ε, ε, αυτή την υποχρέωση και γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. όλα τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα θεσμικά όργανα όταν αποφασίζουν για το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα παραμελούνται πλήρως από τα θεσμικά όργανα. Βασίζονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 και τα θεσμικά όργανα δεν ε, συμμορφούνται με τις αποφάσεις ε, που θα μας έδιναν ε, το δικαίωμα πρόσβαση σε έγγραφα. Με την αναδιατύπωση λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να ευθυγραμμίσουμε τον κανονισμό με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε να βασίζεται σε αυτόν τον κανονισμό και δεν θα επιτρέπει πλέον η κατάσταση στα ευρωπαϊκά όργανα να αγνοούν ή να παραμελούν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντική ευκαιρία αυτή η αναδιατύπωση για να συμμορφωθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σύμβαση του Όρχους και για να εφαρμόζεται καλύτερο ο κανονισμός από τα θεσμικά όργανα της κοινότητας. Για τη σωστή εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θέλουμε να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογή του δικαιώματο πρόσβαση στα έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναής. Με τη δική σου παρέμβαση ξεκίνησε αυτή η κατηγορία των οργανώσεων και προσώπων που δοκίμασαν ε, τους κανόνες αποφάσεις του δικαστηρίου ε, και ενσωχάσει του δικαστηρίου και τη δημοσιολαβητή βελτιώθηκε η πρόσβαση στα έγγραφα και στην ενημέρωση. Και ελπίζουμε ότι τώρα η νομοθεσία θα ε, καλύψει τα κενά, ώστε δεν θα πρέπει να χρονοτριβεί ο κόσμο για να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Εν αυτή τη ενία είναι εκατό να γνωρίζουμε ότι συνήγορο του πολίτη παρέχει τι υπηρεσίε του δωρεάν. Α συνεχίσουμε με τα χαρά. δίνω το λόγο στον Άνε Κένιγκ που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων από την Σουηδία, θα αναφερθεί στα στις και τη βελτίωση της καταστάσεω πλευράς των, επαγγελματικών, των επαγγελματιών χρηστών του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Φοβούμαι ότι δεν θα τηρήσω ακριβώς τη γραμμή που ορίζει το θέμα. Θέλω να επεκταθώ λιγάκι. Χαίρομαι που ήδη αναφέρθηκε δύο φορές η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά την ελευθερία της ενημέρωσης εν γέννη. Διότι τώρα βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή μας Ομοσπονδία που καλύπτει περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες και 250.000 μέλη στην Ευρώπη ότι η διάδοση των πληροφοριών το απόθεμα πληροφοριών του ΣΥΠΗΝ όλο και μικραίνει. Οπότε η πρόσβαση στα έγγραφα είναι κρισίμου σημασία και για τους δημοσιογράφους και για τους άλλους πολίτες και θα ήθελα να θέσω το ευρύτερο πλαίσιο όπου διαβλέπουμε πολλά προβλήματα. Φερρυπίν σε μερικούς μήνες θα παρα, παρατηρούμε ότι πέρασε η δεκαετία μετά τα γεγονότα της 11 η Σεπτεμβρίου. Οι τρομοκρατικές πράξεις ε, στις ΗΠΑ ακολουθήθηκαν από σειρά νομοθεσιών ε, αντιτρομοκρατικών στο Ρέικιαβικ, Ισλανδία, υιοθετήθηκαν κανόνες το 2009, έχουμε τη διακήρυξη του Ρέικιαβικ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εκεί αναφέρεται σαφώς ότι εκείνοι που υπέγραψαν το, τη διακήρυξη πιστεύουν ότι προχωρήσαν πάρα πολύ μακριά όσον αφορά ε, τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης ότι θα πρέπει οι τρομοκρατικοί νόμοι να αναθεωρηθούν και όλη η εθνική νομοθεσία να αναθεωρείται ετησίω σύμφωνα με τη σύσταση αυτή που υιοθετήθηκε. Και στόχο είναι να επιστρέψουμε στην πορεία μα όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωση και των δημοσιογράφων. Από ό,τι γνωρίζω, καμία χώρα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, κανένα μέρο του Συμβουλίου τη Ευρώπη και επίση μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώση που πολλέ περιπτώσει δεν ξεκίνησαν τη διαδικασία. Τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συνεχίζουν με την κράτηση στοιχείων έλεγχο, ε, παρακολουθούν τις επικοινωνίες μέσω τηλεφώνου και υπολογιστών ε, και είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον να ε, προστατεύουν τις πηγές τους δημοσιογράφοι. Το κλίμα για τα μέσα ενημέρωσης γίνεται όλο και πιο κλειστό. Αντιθέτως, δεν επικρατεί άνοιχτη προσέγγιση. Έχουμε το βρετανικό παράδειγμα. Επαγγελματική χρήση των φωτογραφιών εμποδίζεται από την αστυνομία. Εμποδίζονται οι φωτογράφοι να καλύψουν διαδηλώσει και άλλε εκδηλώσει και από τι υποψήφιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώση, όπω στην Τουρκία, περίπου 70 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι γιατί έκαναν τη δουλειά του, αναφέροντα τα γεγονότα. Συνάντησα τον πρόεδρο τη Ένωση Δημοσιογράφων στην Τουρκία, τον Ατσάνι Πέσκη, τι προάλλε και μου είπε ότι υπάρχει ένα κλίμα φόβου που επικρατεί μεταξύ των δημοσιογράφων διότι πολλοί δημοσιογράφοι ε, δέχονται απειλές ε, μέσω ταχυδρομείου και μέσω τηλεφωνημάτων. Η πρόσβαση λοιπόν στα έγγραφα θα πρέπει να ειδωθεί από αυτή την οπτική γωνία, δηλαδή το κλίμα επικρατεί που είναι λιγότερο ανοιχτό, λιγότερη ελευθερία για τα μέσα ενημέρωσης και για, τα... για τους δημοσιογράφους τα ΜΜΕ και πολλοί δημοσιογράφοι σε πολλά κράτη-μέλη λόγω των εθνικών νόμων έχουν προβλήματα να κάνουν τη δουλειά του. Το πρόσφατο παράδειγμα βεβαίω είναι νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία και εμεί τοποθετηθήκαμε όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, κάθετα κατά αυτού του νόμου, αλλά είδαν πολλές ευρωπαϊκές, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι λείπει ποιοτική ενημέρωση των πολιτών για εμπορικούς λόγους, ε, επειδή τα μέσα ενημέρωση, ε, λόγω συγκέντρωση των μέσων ενημέρωση, ο δημόσιο τομέα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, λόγω εθνική νομοθεσία, διότι υπάρχει έλλειψη κατανόηση από πλευρά κυβερνήσεων, στον φάρ την ανάγκη που υπάρχει να παρέχεται δημοσιογραφική πληροφορία σε δημόσια αγαθό. Ε, η δημοσιογραφία έχει ένα σημαντικό εργαλείο στη δημοκρατική διαδικασία. Λοιπόν, οι κανόνε είναι χρήσιμοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόσβαση ε, στι πληροφορίε. Ήταν χρήσιμοι, είδαμε ε, βοήθεια το δικαστήριο, τι αποφάσει του δικαστηρίου, όμω δυστυχώ είδαμε κάποια άλλα παραδείγματα που το δικαστήριο του Ευρωπαϊκού αποφάσισε προ την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, το 2008 ένα Σουηδό δημοσιογράφο προσπάθησε να έχει πρόσβαση σε έγγραφα όσον αφορά καταγγελίε για τον ανταγωνισμού στον τομέα των επιδοτήσεων προ τα μέσα ενημέρωση ε, η όλη εκδίκαση υποθέσεω ήταν ανησυχητική. Το επιχείρημα για να μην δοθούν τα έγγραφα τελικά ήταν ότι δεν ήταν προ το όφελο του κοινού η υπόθεση. Και αυτό με το ιστορικό ζωή συζητήσει που έλαβε χώρα στη Σουηδία όσον αφορά το σύστημα των επιδοτήσεων και τι δυνατότητε να παραμείνει ένα σύστημα με παραπάνω από μία πρωινή εφημερίδα σε δύο μεγάλε πόλει τη ε, χώρα. Ο Στέφαν Ντόλεφ, επίση κατά τη διάρκεια τη διοίκη, ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόβλημα ήταν πολύ ευαίσθητο ε, θα έπρεπε το αίτημά του η πρόσβαση στα έγγραφα να περιμένει. Παραπάνω από τι 15 μέρε που προβλεπόταν, χωρί κανένα δισταγμό δόθηκε αυτή η απάντηση λοιπόν. Για του δημοσιογράφου που ζουν στην ψηφιακή εποχή, στην πραγματικότητα έχουμε προθεσμία κάθε δευτερόλεπτο. Ε, και λόγω και του διαδικτύου βεβαίω. Ήδη 15 μέρε είναι εξαιρετικά μακρά περίοδο να πρέπει να περιμένουμε για την παροχή των πληροφοριών. Ε, Επίση, σχετικά με τι επιδοτήσει ε, στου γεωργού αυτή τη φορά, αποφασίστηκε πέρσι ότι ε, εκατομμύρια χρημάτων των φορολογουμένων πηγαίνουν σε, σε άτομα ή σε μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς να δίδονται πληροφορίες που χορηγούνται και δεν μπορούν να αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές για τις επιδοτήσεις στις ιστοσελίδες. Και το ίδιο στους αποδέχτες στους Ιδούς ε, των επιδοτήσεων οι πληροφορίες μέσω του νόμου για ελεύθερη ενημέρωση διατίθεται πληροφορίες η ακαιρεότητα των μέσων ενημέρωση φαίνεται ότι θεωρείται λιγότερο σημαντική από τι ανάγκε του φορολογουμένου για να βλέπει πώ χρησιμοποιούν τα χρήματά του. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναθεώρηση του κανονισμού για ανοιχτή προσέγγιση και την ευθυγράμμιση του με τι συνθήκε τη Λισαβόνα συμπεριλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη και αν γίνει αυτό θα είναι ένα βήμα πρόοδου. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καλύπτουν και την πορεία των εθνικών φορέων οι αναθεωρημένοι κανόνε ανοιχτή προσεγγίσεω τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των θεσμικών οργάνων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περίπλοκου κανόνε όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα και κατηγορίε εγγράφων. Είναι κρίσιμο σημασία να μην υπονομεύεται ό,τι ήδη υπάρχει όσον αφορά του κανόνε. Αλλά βεβαίω ίσω θα είναι. Είμαι ένα από του λίγου εδώ, ελπίζω όχι, που ασχολούμαι με το θέμα. Όταν εσεί στο Κοινοβούλιο συνεχίζετε σημαντική σα εργασία για την ανοιχτή προσέγγιση, εξετάστε το αυτό στο πλαίσιο που προσπάθησα να, να σα παρουσιάσω και όπως αφορά τις αντιδράσεις στο Wikileaks ή Brussels, Leaks. Χρειάζεται ένα σύστημα ανοιχτό, και, αλλά το ανοιχτό πρέπει να δίνει αποτελέσματα. Ε, διότι υπάρχουν νέοι τρόποι ε, παρουσίαση των πληροφοριών σε ευρία κλίμακα, που όλες οι πληροφορίες κανονικά θα πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ανοιχτά στο ευρύ κοινό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κένινγκ, ιδιαίτερα για την έκκλησή σας να μην ξεχάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο σε θέματα ασφάλεια, κρατικής ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας που ε, αποτελούν πλέον πρόσκομα ε, και στην πρόσβαση στην πληροφορία γενικά του κοινού αλλά και ιδιαίτερα των δημοσιογράφων και άλλων οργανώσεων που προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και ιδιαίτερα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, ελευθερίας έκφρασης. Τώρα περνάω στον Τόνι Μπάνιαν. Κάτι θα ξέρει παραπάνω για τα Brussels Leaks. και πώς ολόκληρες ε, κατηγορίες ε, εγγράφων αποκρύπτονται ε, και δεσμεύονται έτσι ώστε να μην δημοσιοποιηθούν. Τόνι. Ο Τόνι αντιπροσωπεύει την State Watch. Ευχαριστώ. Θα είμαι θετικός για το πώς η προσαρμογή του κανονισμού στη Συνδίκη της Αβώνας μας δίνει ευκαιρία να ανοίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο αρχικός κώδικας πρόσβασης είχε εγκριθεί το 1993, ε, υπήρχαν μόνο δύο εξαιρέσεις στον κώδικα. Στο άρθρο 4.1 και στο άρθρο 4.2, ε, που αντιστοιχούν στο 4.1 και 4.2 του κανονισμού, του σημερινού κανονισμού. Όταν ε, ήρθε το συνδίκτο Άμστερνταμ, εισήχθη μία ακόμα κατηγορία που την πρότεινε η Κομισιόν η Κομισιόν έλεγε έπρεπε να αποφύγουμε ε, παρεμβάσεις στην διαδικασία λήψη αποφάσεως και τη πρόορη δημοσιοποίηση εγγράφων που θα οδηγούσε σε παραπλάνηση. Όταν η δημοσιοποίηση επηρεάζει την διαδικασία λήψη αποφάσεως, τα έγγραφα δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, έλεγε η Κομισιόν. Ε, δηλαδή ήθελε να προστατέψει ε, το χώρο σκέψης των υπαλλήλων της. Ε, η ίδια απαγόρευση μπορεί να ισχύει και μετά τη λήψη όμω αποφάσεων, αν αυτή η δημοσιοποίηση θα επηρέαζε μια μελλοντική λήψη αποφάσεων. Οπότε, πέραν των γενικών εξαιρέσεων, προσθέθηκε και αυτή η τρίτη εξαίρεση περί παρέμβαση στην διαδικασία λήψη αποφάσεων θεσμικών οργάνων. Η ε, ετήσια εκθέση του 2009 αναφέρει ότι το 25% των αιτήσεων Ε, που απορρίπτονται, απορρίπτονται με βάση το άρθρο 4.3. Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών προσπαθούσε να μάθει τι συζητείται στα θεσμικά όργανα, τι θα νομοθετηθεί. Το επιχείρημα είναι ότι όταν συζητούν οι νομοθέτες θα πρέπει τα έγγραφα τα οποία συζητούν να είναι δημόσια. Αυτό είναι κανόνα οποιασδήποτε δημοκρατία. Και τι σημαίνει στην πράξη. Σημαίνει ότι όταν ε, συναντά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι επιτροπέ του, όλα τα έγγραφά του είναι δημόσια. Όταν όμως, ε, και όταν το Συμβούλιο ε, συναντιέται, συνέρχεται νομοθετικά, θα πρέπει επίσης να συμβαίνει το ίδιο, αλλά δεν συμβαίνει. Το ίδιο και στην Κομισιόν. Στην Επιτροπή Λίμπε, λοιπόν, το 2008 και 2009 το 84% των μέτρων που εγκρίθηκαν, εγκρίθηκαν σε κλειστέ και σε συναντήσει που έγιναν και κλεισμένων των θυρών. Οπότε, οποιαδήποτε δημοκρατία σέβεται τον εαυτό τη, θα πρέπει να έχει μια ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών που θα ε, συμμετέχει στη συζήτηση και θα παρεμβαίνει. Η πρόταση Κομισιόν για τροποποίηση του κανονισμού, έτσι ώστε να, προσαρμοστεί στη Λισαβόνα, μα δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούμε από το άρθρο 4.3. Η Κομισιόν από την άλλη μεριά πιστεύει ότι αυτή η διαδικασία σημαίνει απλώς τη διεύρυνση των οργάνων τα οποία καλύπτονται. Όμως, στο άρθρο 15.3, ε, παράγραφος 5, η συνδίκη Λισαβόνας λέει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να δημοσιεύουν όλα τα έγγραφα σχετικά με τις ε, νομοθετικές διαδικασίες. Πιο καθαρό από αυτό δεν μπορεί να είναι. Επίσης το άρθρο 11.1 λέει απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση, να δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες και σε οργανώσεις τους να, δίνουν τη γνώμη τους για οποιαδήποτε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα δουν την άποψή τους και τη γνώμη τους άμα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Και υπάρχει άλλος ένας λόγος για την απαλυφή του 4-3. Το 4-3 βασιζόταν στο Άμστερνταμ. Είχε νομική βάση το Άμστερνταμ. Δεν υπάρχει πλέον νομική βάση στη Λισαβόνα για την, ε, σοβαρή, ε, ε προστασία της πληροφορίας. Συνεπώς, το 4-3 δεν έχει βάση τη συνθήκη πλέον. Η συνθήκη Λισαβόνα θα μπορούσε να είναι πιο σαφή. Λέει ότι τα έγγραφα, τα σχετικά με τη, με τις διαδικασίες, η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια τη διαδικασίας, όχι μετά. Και άλλωστε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα το ανέφερε το 2010. Δεν είναι δυνατόν ε, η ανοιχτή προσέγγιση να παγιώνεται από την συνθήκη αλλά να μην αντικατοπτρίζεται αυτό στο κανονισμό. Το 1999, θυμάμαι, ο κ. Σότμαν είχε πει ότι, ότι ε, υπήρχαν ε, δεινόσαυροι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο που ήθελαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και εξακολουθούν να υπάρχουν. Ε, μετά το 2001 ε, ε, είχαμε τη, αποκτήσαμε το 50% αυτό που θέλαμε. Δεν θέλουμε αυτό να περιοριστεί. Έχουν, έχει δικαίωμα η κοινωνία των πολιτών να ξέρει τι συμβαίνει και η, συνοθεία, και η συνθήκη της Λισαβόνα μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξαναβάλουμε τους δεινόσαυρους πίσω στην τουλάπα από την οποία είχαν βγει. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, χρήσιμο το ότι αναφέρατε το έργο του κυρίου Σάντεμαν. Ε, είχαμε δύο εξαιρετικού διαμεσολαβητέ ε, που τόνισαν το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν. Ίσως η εξαίρεση 4.3 είναι κάτι που χρησιμοποιείται ευρύτατα και είναι κατά του πνεύματος, ε, του ανοιχτού πνεύματος, του ότι πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν και να ενημερώνονται. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον Ιβ Στάινιτς να λάβει το λόγο, να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό χώρο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κοινή γλώσσα. Ο κ. Στάινιτς ε, είναι διευθυντής στη Διεύθυνση ΓΑΜΑ από την Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές που μου δίνουν τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουν συντομία τη δουλειά που κάνουμε για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα νομοθετικά κείμενα. Καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η δική μου παρουσίαση θα είναι πάρα πολύ στεγνή, τεχνική και χωρίς ε, ενδεχομένως μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας πω καταρχήν ποια είναι η εντολή που μας έχουν δώσει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα σας παρουσιάσω καταρχήν αυτό το οποίο βλέπουν οι χρήστες. Έχουμε ένα σημείο ανοιχτής πρόσβασης και από πίσω υπάρχουν και αυτά τα οποία δεν βλέπουν οι χρήστες, όλο το σύστημα πληροφορικής το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτό το οποίο βλέπουν οι χρήστες. καθώς επίσης και τη μοντελοποίηση και την προτυποποίηση που μας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τη διαχείριση γνώσης και για τις ε, χρήσεις του διαδικτύου και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δημόσια δεδομένα. Ο κύριος Μπερνάρ Μπονζόν από το Εθνικό Συνδικάτο στη Γαλλία έγραψε το 2004 ότι όλοι οι συντάκτες και εκδότες θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κοινά πρότυπα σχετικά με το περιεχόμενο ούτω ώστε να υποφελούνται όλοι οι χρήστες των νομικών βάσεων δεδομένων. Επτά χρόνια αργότερα έχουμε τώρα ένα κοινό χώρο όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη μια κοινή γλώσσα, ενώ ο κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε στον πολίτη εύκολη πρόσβαση στα νομοθετικά κείμενα και διαφάνεια. Αυτό δεν σημαίνει η δυνατότητα πρόσβασης στα νομοθετικά κείμενα δεν σημαίνει μόνο να είναι διαθέσιμα τα έγγραφα, σημαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν τα έγγραφα μέσα στο νομικό και θεματικό τους και διαδικαστικό τους πλαίσιο. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για ανοιχτή πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτό πρέπει να γίνεται μέσω μιας ε, ε, δικτυακής, ε, κοινής δικτυακής πύλης. χρησιμοποιούμε την προτυποποίηση στα συστήματα πληροφορικής και χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά. Η προτυποποίηση σημαίνει μοντελοποίηση των δεδομένων και των διαδικασιών με προτυποποιημένη χρήση κωδικών Ε, και υπάρχουν συγκεκριμένοι πίνακες όπου είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο, το κείμενο. Uh, <clears throat> το, το σημείο κοινή πρόσβαση είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Κάπω έτσι εμφανίζεται, όπω αυτό που είναι στην οθόνη και ίσω πολλοί από εσά το γνωρίζετε αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Είναι παιδεία στα οποία μπορείτε να μπείτε και να κάνετε αναζήτηση όλων των τομέων και όλου του περιεχομένου το οποίο διαθέτουμε. Έχουμε ένα γενικό μοντέλο και κάποιες ε, επιμέρους πτυχές, αυτά που βλέπετε ε, στο αριστερό τμήμα της οθόνης, με περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες, τον τύπο του εγγράφου κλπ. Και δίνοντας αυτές τις επιμέρους πτυχές, προσφέρουμε στο χρήστη δυνατότητα ε, να έχει πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεσμάτων. Και οι περισσότερο πεπειραμένοι χρήστες που μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν πολύπλοκα νομικά, ε, νομικές ιστοσελίδες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο EUR-LEX που έχει περισσότερες δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης. για να σας εξηγήσω τι εννοώ όταν σας είπα ότι πρέπει να δίνουμε το έγγραφο μέσα στο σωστό του πλαίσιο. Εδώ βλέπουμε την νομοθετική διαδικασία, παρουσιάζονται τα έγγραφα με τη χρονική σειρά και με την ακολουθία γεγονότων που οδήγησαν στη διαμόρφωση του τελευταίου εγγράφου. Αυτά όσον αφορά αυτό που βλέπουν οι χρήστες, το front end. Ας δούμε τώρα και αυτά τα οποία ε, δεν βλέπουν οι χρήστες. Υπάρχει το σημείο κοινή πρόσβασης, ε, οι μηχανές αναζήτησης και οι δείκτες. Τα περιγραφικά μεταδεδομένα είναι απόλυτα απαραίτητα και η καρδιά του συστήματος βρίσκεται κάτω από το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα κοινά δεδομένα. Αυτοί οι δύο κύκλοι που έχετε δεξιά με το κίτρινο και πράσινο χρώμα, το πρόγραμμα ε, Record και το πρόγραμμα Eurovoc είναι προγράμματα τα οποία αφορούν το αρχείο μεταδεδομένων όπου έχουμε όλα τα τυποποιημένα μεταδεδομένα στο Record και στο Eurovoc έχουμε ένα πολύγλωσσο θησαυρό υλικού. Εδώ βλέπετε τη μοντελοποίηση των δεδομένων, παρότι δεν μπορείτε να το δείτε πολύ καλά γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα στην οθόνη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εδώ έχουμε μια διαδικασία. Η διαδικασία ορίζεται από κάποια σετ μεταδεδομένων και η διαδικασία συμπεριλαμβάνει και κάποια ε, γεγονότα με συγκεκριμένο έργο το οποίο περιλαμβάνεται και με συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δηλώσεις. εκφράζεται το έργο στις διάφορες γλώσσες και η εμφάνισή του γίνεται σε αρχείο PDF. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα παράδειγμα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Επέλεξα ένα παράδειγμα. το οποίο θεωρώ ότι θα σας είναι περισσότερο οικείο γιατί αφορά κάποιους κωδικούς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν τέσσερις τέτοιοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό περιβάλλον και που οδηγούν στο ίδιο σετ εγγράφων. Αποφασίσαμε λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο κωδικό με τις προϋποθέσεις χρήσης και το περιεχόμενο το οποίο τελικά θα έχουμε σε κάθε μία από τις 23 γλώσσες. Είναι τεράστιο το έργο προτυποποίησης αυτών των μεταδεδομένων. Με κίτρινο χρώμα βλέπετε αυτό το οποίο έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Με ροζ χρώμα είναι το έργο το οποίο ακόμη βρίσκεται να εξελίξει. Συνεργάζονται όλα τα θεσμικά όργανα στην προσπάθεια αυτή. Ένα σχόλιο της Προέδρου εκτός μικροφώνου. Είναι πολύ ε, ε, δύσκολο το έργο το, της συνένωσης των μεταδεδομένων. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και περνώ λοιπόν στην σύνοψη της παρουσίασής μου. Χρειαζόμαστε ποιότητα και ποιότητα σημαίνει ακρίβεια όσον αφορά την αξία των μεταδεδομένων και ε, εξού και είναι σημαντική η χρήση βιβλιογραφίας και νομικών δικτών. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνεπή τρόπο τα πρότυπα για την παρουσίαση και μεταβίβαση και αποθήκευση δεδομένων. Τα πρότυπα αυτά πρέπει ε, να υιοθετούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πιο εύκολη επικοινωνία και νέα χρήση των εγγράφων, επακριβή ερμηνεία των σχετικών μεταδεδομένων και θα αποφεύγονται παρανοήσεις καθώς και απώλεια χρόνου. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η προτυποποίηση των μεταδεδομένων δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης περιεχομένου από πολλές πηγές, από ένα σημείο πρόσβασης ή από μια διαδικτυακή πύλη. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και αν θέλετε κάποιε διευκρινήσει για να κατανοήσετε καλύτερα την παρουσίασή μου, θα είμαι στη διάθεσή σα. Αυτό που προσπαθείτε να δημιουργήσετε είναι όνειρο για μας. Δηλαδή, κατάσταση όπου έχουν εύκολη πρόσβαση πολίτες πληροφορίες. Διερωτώ με μήπως χρειάζεται πάνελ καταναλωτών για να δοκιμάσουν οι τελικοί χρήστες πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε 10 λεπτά, ένα τέταρτο για ανταλλαγή σχολείων, υποβολή ερωτήσεων, υποβολή απαντήσεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας ακούσουμε τους σημερινούς ομίλητες. Και τα μέλη του Κοινοβουλίου βέβαια. Η κυρία Μόρβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την άκρο ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση. Είμαι νομικός από την Ουγγαρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανεξάρτητο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα νομίζω ότι μιλάμε για την βάση, τα βασικά, πολύ βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είμαι πολύ απογοητευμένη που δεν είναι παρόντα περισσότερα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Θυμήθηκα τον πατέρα μου σήμερα δύο μήνες μετά την πτώση του κομμουνισμού στη χώρα μου. Όταν είπε ότι είναι φρικτό αυτό που συνέβη. Στην τηλεόραση ανακοίνωσαν μόλις τώρα ότι ένα δημόσιο έγγραφο θεωρείται ως απόρριτο από την ελεύθερα εκλεγμένη κυβέρνηση, την πρώτη μετά από 30 χρόνια. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έγινε βασική αλλαγή του συστήματος. Γιατί πράγμα μιλάμε τώρα. Μιλάμε για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες της δημοκρατίας. Στην πραγματική δημοκρατία πιστεύω ότι όλη η εξουσία που έχει η κυβέρνηση προέρχεται άμεσα ή έμεσα από το λαό και ο λαός έχει το δικαίωμα να ελέγχει και να υποπτεύει αυτά που κάνει η κυβέρνηση εκ μέρους του. Σε μια δικτατορία ή ήμι δικτατορία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η κυβέρνηση έχει όλη την εξουσία. Μια ελίτ έχει την εξουσία και η αδίποτε εξουσία του ατόμου του δίδεται ή της δίδεται από την κυβέρνηση. Εντελώς διαφορετικές ερμηνείες. Και αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το βασικό νόημα, το θεμελιώδες νόημα της δημοκρατίας. Ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να καταλάβει ή πολίτης ότι ελέγχει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Διότι όλη η εξουσία θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προέρχεται από εκείνη. Γι' αυτό είναι θεμελιώδες αυτό που συζητούμε. Και το ερώτημα μου, ζητώ που μακρηγόρησα, αλλά ενθουσιάζομαι, ξέρετε, με αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά, πολύ θεμελιώδη. Κυρίως Απευθύνομαι προ τον δικηγόρο συνάδελφο. Θα χρησιμοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το σύστημα αυτό, θα προσφύγετε στο Στρασβούργο τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει τη σύμβαση. Διακόπτει η Πρόεδρος και δεν ακούμε τη συνέχεια της παρεμβάσεως, γιατί μιλάνε και οι δύο μαζί. Λοιπόν, υπήρξαν παρεμβάσεις από και θα υπάρξουν παρεμβάσει και από το πάνελ, από τους ευρωβουλευτέ. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Διαμαντούρο, έχετε το λόγο. Ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά την πολύ σημαντική παρουσίαση του κυρίου Στάινιτ. Αυτό που προσπάθησε να μας δείξει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά πάει στην καρδιά του αναγκαίου. Να κάνω μια φιλική σύσταση πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μεταφράζετε τα πολύ στεγνά στοιχεία σε μια παρουσίαση που θα είναι πιο εύληπτη για τους χρήστες. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ξέρω από τη δική μου δουλειά. Χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες αλλά πολλά εξαρτώνται από την ικανότητα που έχουν τα θεσμικά όργανα, οι φορεί να κάνουν αυτά όλε τι πληροφορίε πιο ευκολοχώνευτε, πιο εύληπτε. Τα στοιχεία είναι πολύ στεγνά από τη φύση του. Δεν σα δίνω μια λύση. Σα δίνω μια φιλική σύσταση και ενθουσιώδη υποστήριξη για αυτά που προσπαθείτε να κάνετε και ελπίζω να βρείτε μια λύση. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπράουερ έχει το λόγο. Καταρχάς, σας συγχαίρω για τη διοργάνωση της ακρόασης. Είναι πολύ καλό που συζητούμε την αιχτή προσέγγιση και τη διαφάνεια σήμερα. Έχω ένα ερώτημα. Ίσως απευθυνόμενος προς τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή και ίσως απευθυνόμενο σε μερικούς από εσά που ασχολείστε με την αναθεώρηση του κανονισμού 1049. Ερώτηση λοιπόν. Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε την υπερβολική ταξινόμηση των στοιχείων Πολύ συχνά ταξινομούνται τα έγγραφα, θεωρούνται περιορισμένης ε, διάδοσης, εμπιστευτικά, απόρριτα κλπ. Και καμιά φορά αυτό δεν δικαιολογείται. Είναι πολύ σημαντικό και πήγον ζήτημα, αλλά ε, δυσεπίλητο. Και για τα δικαστήρια. Ποια είναι η ιδεώδης κατάσταση, ότι δεν χρειάζεται να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο ότι έχει κανείς ε, μπροστά του ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να προσφύγει. Αλλά τότε είναι που τίθεται το θέμα της ταξινομήσεως και του χαρακτηρισμού των εγγράφων. Ναι, λέει η Πρόεδρος, είναι βασικό θέμα αυτό για τις συζητήσεις μας. Ελπίζω να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις σε αυτό. Να ξεκινήσουμε από το διαμεσολαβητή και μετά πάμε στον Μάικλ Κάσμας και στον Τόνι Μπάνιον και μετά θα δώσω το λόγο και στην ε, Αναίδα για να δώσει απάντηση στην ερώτηση της ε, δικηγόρου από την Ουγγαρία. Θα είμαι σύντομο, λέει ο κ. Θα δώσω μερική απάντηση που αφορά το διαμεσολαβητή. Το συνήγορο του πολίτη. Εγώ δεν μπορώ να πω πώ κατηγοροποιούνται τα έγγραφα. Αυτά είναι αποφάσει των θεσμικών οργάνων. Εγώ ασχολούμαι με την εκτέλεση των αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, Τροποποιήθηκε και, τα, η δική μου δικαιοδοσία το 2008, η εξουσία μου, ε, χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων και τώρα έχω πρόσβαση σε κάθε είδους ε, στοιχείο και σε όλα τα έγγραφα ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους και το βαθμό εμπιστευτικότητας. Τι περιορισμό έχω. Ε, πρέπει να έρθω σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο πριν έχω την πρόσβαση ε, του όρου υπό του οποίου θα έχω την πρόσβαση. Το δοκιμάσαμε ήδη αυτό μια φορά κατά τη διάρκεια τη Σουηδική Προεδρία και θέλω να χαιρετήσω την ενθάρρυνση τη Σουηδική Προεδρία και μπόρεσα να πείσω το Συμβούλιο να θεσπίσει κάποιους κανόνες για να επιτρέψει την πρόσβαση στα λιγότερα διαβασμισμένα έγγραφα, τα περιορισμένης διάδοσης, τα αριστρά ο συνήγορος του πολίτη έχει πρόσβαση τώρα. Έχουμε ένα, ένα καλό προηγούμενο και έτσι υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Δεν απαντώ στο ερώτημά σας, δεν έχω την εξουσία εγώ να καθορίσω τι είναι διαβαθμισμένο, πώς είναι διαβαθμισμένο. Απλώς μπορώ να αποφασίσω πώς μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ, ο Μάικλ. Ευχαριστώ, Χάιντι. καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Μοβάη για το πάθος που έδειξε για τις πληροφορίες και την πρόσβαση σε αυτές, διότι πραγματικά είναι κάτι που ενισχύει τη δημοκρατία. Και βεβαίω υπάρχουν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ζήσει υπό δικτατορίε. Άρα υπάρχει μια πραγματική εμπειρία όσον αφορά την στέρηση τη δημοκρατία. Ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υπερβολική διαβάθμιση των εγγράφων έχουμε κοινού κανόνε για τα θεσμικά όργανα και για όλου του φορεί και αυτοί και είναι οι κανόνε για τη διαβάθμιση των εγγράφων θα πρέπει να δημοσιεύονται. Είναι εσωτερικοί κανόνε που δημοσιεύονται και τότε αυτή η διαβάθμιση μπορεί να αμφισβητηθεί. Και αυτή είναι η προσέγγιση που ακολούθησε μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού 1049. Ευχαριστώ, Μάικλ. Ο Τόνι έχει το λόγο. Δύο πράγματα να πω, λέει ο κ. Μπάνιον. Υπάρχει και άλλο ένα επίπεδο μερική πρόσβαση και σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από τον ε, υπάλληλο που ασχολείται με το έγγραφο. Για τα διαβασμένα έγγραφα είναι ευρύτερο τομέα. Αυξάνονται οι αριθμοί των εγγράφων που είναι διαβαθμισμένα στο Συμβούλιο. Υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, για προστασία των δεδομένων που αφορά την ιδιωτική ζωή των ατόμων ε, για κάθε έγκλημα ανηλίκου κλπ. Πρέπει να δούμε τι διαπραγματεύονται εκ μέρου μα. Γιατί κάποια αναβαθμίζεται ε, η πιστευτικός χαρακτήρας κάποιων εγγράφων με ποια απόφαση. Πρέπει να δούμε πώ συζητείτε το θέμα, ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθείτε και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ο Μάικλ θέλει να δευτερολογήσει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα έγγραφο που ελπίζω ότι είναι δημόσια διαθέσιμο γιατί πιστεύουμε στη διαφάνεια και στην ανοιχτή προσέγγιση και σελίδα 21 εισάγουμε την έννοια της διαβαθμίσεως των εγγράφων χρησιμοποιήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου δεν υπονομεύουμε την ε, αρχή της ταξινόμησης και της διαβάθμισης όπου αυτό απαιτείται και έχουμε λοιπόν τη διαβάθμιση και μετά λεπτομερώς περιγράφουμε γιατί έχει αυτό το χαρακτηρισμό αυτό το έγγραφο. Άκρος απόρριτο Φερρυπίν. Αυτό είναι κάτι που ισχύει για πληροφορίες και υλικό η αποκάλυψη του οποίου θα δημιουργούσε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω ή για ένα ή περισσότερα από τα κράτη-μέλη της Ενώσεω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να πούμε, μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαβάθμιση εάν το έγγραφο ε, καλύπτεται από, από αυτόν τον κανόνα και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε τελικά τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την ταξινόμηση που ε, ακολουθείτε. Ευχαριστώ. Ε, η ανησυχία που έχουμε είναι η εξή. Υπερβολική διαβάθμιση ταξινόμηση, να γίνονται πιο πολλά απόρριτα έγγραφα από ό,τι χρειάζεται και ότι δεν εφαρμόζονται κανόνε και έχουμε έγγραφα μπροστά μα στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο. Και τίθεται το ερώτημα, ποιο ελέγχει το πώ διαβαθμίζονται τα έγγραφα και πώ μπορούμε εύκολα να το συζητήσουμε αυτό για την κατηγοριοποίηση και το χαρακτηρισμό που δίδεται σε συγκεκριμένο έγγραφο. Αν επιτρέπετε, λέει ο κύριος Κάσμαν, ο Νικηφόρος το ανέφερε. Και αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αυτή που αναφέρθηκε. Και αυτό θα είναι ε, κάτι το οποίο θα το αναλάβει ο αρμόδιος για την ε, ενημέρωση και τη χορήγηση πληροφοριών, η πρόεδρος. Να πω ότι όταν ε, θεσπίστηκε ο κανονισμός, κάποιοι εμπειρογνώμονες είπαν, είπε ότι είναι σαν ματριός καροσική, σαν το κουκλάκι το ξύλινο. Ανοίγει λοιπόν το έξω κουκλάκι και έχει νέο κουκλάκι πιο μέσα και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος θα έπρεπε να επικρατεί και μετά έχουμε το άρθρο 9 του κανονισμού για τα ευαίσθητα έγγραφα ε, που θεωρήσαμε απογοητευτικό συμβιβασμό τότε. Και έχουμε και του εταιρικού κανονισμού και του κανονισμού για τη διαβάθμιση κλπ. Και, και αυτό που προσπαθεί να πει ο Μάικλ Κάσμαν με το σχέδιο έκθεσή του για την αναδιατύπωση είναι ότι όλα πρέπει να τεθούν σε ένα ενίο πλαίσιο. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πιστεύω να το σκεφτούμε. Ε, ορίστε, Νικηφόρα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι κάτι που πρέπει να πούμε ξεκάθαρα. Ακριβή διατύπωση. Η σωστή γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε εγγυημένη πρόσβαση. Ακριβής διατύπωση. Τι είναι προσβάσιμο, τι δεν είναι προσβάσιμο ούτως ώστε να περιοριστούν οι φαίες που επιτρέπουν καταχρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που ο νομοθέτης θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Από τη στιγμή που σαφώς έχουν καθοριστεί επακριβώς τα όρια, με ακριβή διατύπωση, είναι καλύτερη κατάσταση. Τα δικαστήρια βοηθούν. Τα δικαστήρια διευκρίνησαν πάρα, πολύ, ε, πάρα πολλά αμφίσιμα σημεία, επίμαχα ζητήματα. Η Αναής Μπεχτή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ούτε η αλλω περιμενουμε την αποφαση του ευρωπαικου δικαστηριου ισως θα επρεπε να εχει προσαρμοστει η επιτροπη και το Συμβούλιο με τις αποφάσεις, με την ομολογία ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ας αφήσουμε τις δικαστικές αποφάσεις λοιπόν να πάρουν το δρόμο τους. Ας δούμε τι έχουν ε, να μας πούν αυτές οι αποφάσεις. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν φτάσει μέχρι το δικαστήριο σε πολύ λίγε περιπτώσει. Για μα είναι πολύ καινούριο το ότι καταφεύγουμε στο δικαστήριο. Είναι κάτι νέο και πολύ ενδιαφέρον. Είναι η μόνη περίπτωση στην Ευρώπη που φτάνει μια μη κυβερνητική οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όταν λοιπόν υπάρχει άρνηση πρόσβαση σε έγγραφα, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο δικαστήριο. Σε άλλα θέματα δεν έχουμε δυνατότητα στο δικαστήριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή της Σύμβασης του Όρχους θεώρησε ότι ότι θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί τα ευρωπαϊκά όργανα με αυτή τη διατύπωση και επομένως, είχαμε τη δυνατότητα να ε, καταφύγουμε στο δικαστήριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο του να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά ενδεχομένω θα φτάσουμε και εκεί. Ευχαριστώ. Ε, ε, πρόεδρο, ε, κυρία Χαουτάλα, αυτό που ανέφερε ο κύριος Κιόνιξ στην παρέμβασή του έχουν σχέση με το δικαστήριο του Στρασβούργου. Α συνεχίσουμε τώρα όμως με το δεύτερο τμήμα που ασχολείται με τις προκλήσεις που τίθενται για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα αλλάξουν οι ομιλητές λοιπόν που κάθονται εδώ δίπλα μου στο βήμα και θα ζητήσω καταρχήν από την ε, Helen Derbyshire Τσεσάρε και τον κύριο Σεύκοβιτς να έρθουν κοντά μου εδώ στο βήμα. Okay, yeah, right, yes. Is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. If yeah. you want to break, yeah. if you need to go uh, um, or anything. Uh, uh, um, λοιπόν, όταν ε, ενώ έρχονται εδώ τα μέλη του δεύτερου πάνελ, να σας ενημερώσω για το εξής. Πολλοί από εμά ε, γιορτάζουν την απόφαση του, Ευρωπαϊκού, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την πρόσφατη απόφαση, για την απόφαση πρόσβασης της θέσης των κρατών μελών επί της αναδιατύπωσης του κανονισμού περί ε, κοινής πρόσβασης στα έγγραφα. Και είναι αστείο που τα κράτη-μέλη έχουν τόσα πολλά να κρύψουν για το θέμα της συζήτησης αυτού ακριβώς του ζητήματος της ελεύθερης πρόσβασης. Το δικαστήριο όμως πολύ ρεαλιστικά ε, τους εξήγησε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις των κρατών μελών για το τι πιστεύουν δηλαδή για την αλλαγή των κανόνων, επουδενή ναι, δεν παραβιάζει την ελευθερία των κρατών μελών να αλλάξουν θέση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Το κοινό είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά ότι οι θέσει των κρατών μελών κατά τη διάρκεια τη νομοθετική διαδικασία μπορούν να εξελίσσονται δεδομένη τη γενική συζήτηση, στην οποία πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Ελπίζω να έχω ερμηνεύσει σωστά αυτό το τμήμα τη συζήτηση. Χέλεν, έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Ναι, έχετε, έχετε δίκιο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περίπτωση αυτή που προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά τα οποία βλέπετε στην οθόνη, ότι η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες που θέλουν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν την νομοθετική διαδικασία. Ε, είναι θεμελιώδες. Σε εθνικό επίπεδο, όπως είπαν και άλλοι ομιλητέ, είναι απόλυτα φυσιολογικό να περιμένουμε να γνωρίζουμε τη θέση των πολιτικών κομμάτων και των μελών τη κυβέρνηση. Όλοι οι βουλευτέ, οι υπουργοί που αρνούνται να δηλώσουν δημοσίω τη θέση του για το α ή το β ε, νομοθετικό ζήτημα, ε, δέχονται την επίκριση και του κοινού και ενδεχομένω και, και των μέσων μαζική ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί τι ίδιε ακριβώ προδιαγραφέ ε, δεν είναι μια πολιτική ε, ουδέτερη ζώνη. Ε, μετά την είδηση για την απόφαση του δικαστηρίου, είναι, κάποιος μου είπε εκπλήσωμε που χρειάστηκε να προσφύγετε καν». Είναι ηρωνικό να πρέπει να προσφύγουμε στο δικαστήριο για να αποκτήσουμε γνώση των θέσεων για την αναδιατύπωση του κανόνα για την πρόσβαση, Τον κανόνα για την πρόσβαση είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι ακόμη και τα κράτη-μέλη τείνουν να παραπέμουν στι Βρυξέλλε για αυτά τα ζητήματα. Ζητήσαμε από τι μόνιμε αντιπροσωπείε εδώ στι Βρυξέλλε να μα ενημερώσουν για τη θέση των, του κάθε κράτου μέλου και βλέπετε τι πήραμε. Ένα παράδειγμα αυτό που πήραμε. <laughs> Ένα τέτοιο έγγραφο μα στείλανε. Ε, τελικά βέβαια επαναλάβαμε το αίτημά μας και μας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες, αλλά μόνο 11 από τις 27 χώρες μας έδωσαν τελικά κάποιες πληροφορίες. Και ακόμα και αυτές πολλές φορές μετά από επίμονες οχλήσεις εκ μέρους μας. Για παράδειγμα, κάτω χώρες που φημίζονται για την διαφάνειά τους, στην αρχή αρνήθηκαν ε, να μας απαντήσουν ε, προφασιζόμενοι ε, διεθνείς σχέσεις και μας έδωσαν πληροφορίες μόνο αφού επιμείναμε. Ε, άλλες έξι χώρες αρνήθηκαν επισήμως να μας δώσουν πληροφορίες ε, με δικαιολογία της διεθνής σχέσης ή την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η Γαλλία, είναι πολύ ενδιαφέρον, εφάρμοσε τον κανονισμό 1049 παρόλο ότι το αίτημά μας βασιζόταν στον γαλλικό νόμο του 1978. Οπότε το ρεφλέξ μυστικοπάθεια των Βρυξελών αντικατοπίζονται και σε εθνικό επίπεδο. Άλλε έξι χώρε μα ε, μα είπαν να απευθυνθούμε στην, ε, ε, στο Συμβούλιο. Μας παρέπεμψαν ξανά στο Συμβούλιο. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε Συμβούλιο για να μάθουμε τη θέση τους. Οπότε άντε πάλι πίσω στην αρχή. Οπότε είναι προφανές ότι αν η διαδικασία λήψη αποφάσεων δεν ανοίξει εδώ σε Βρυξέλλες, ε, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν πρόκειται να ανοίξει ούτε καν σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα μπορεί να βλαφθεί η υπάρχουσα πρόσβαση ε, σε εθνικό επίπεδο. Στη δική μας περίπτωση μάλιστα το έγγραφο είχε ήδη διαρρεύσει. Δεν το ξέραμε βέβαια όταν ε, κάναμε την προσφυγή στο δικαστήριο, αλλά κάπου υπήρχε, ε, ακόμη και στο δικό μας site, ε, κρυμμένο. οπότε ε, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Συμβούλιο ε, δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη πίστευε ότι θα προκύψει από δημοσίευση του εγγράφου. Και ε, μάλιστα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο κοινό το δικαστήριο ότι θα καταλάβει το κοινό τις ενδεχόμενες αλλαγές των θέσεων των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ε, το, η ιδέα ότι θα ε, δημιουργούνται προβλήματα στη διαπραγμάτευση με το κάθε κράτος μέλος να τα στυλώνει ε, δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Η ε, διαφάνεια που δεν είναι βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται νόμοι. Ασφαλώς όχι το, ε, μετά την απόφαση του δικαστηρίου άρχισα να λαμβάνω μηνύματα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από παντού σε όλο τον κόσμο. Ε, από την Κένια ένα ακτιβιστή μου είπε ότι αυτή η απόφαση θα ήταν πολύ χρήσιμη για αυτού. Ε, ε, στην Νότιο Αφρική έγινε, δημοσιεύτηκε ένα ολόκληρο άρθρο στο ίντερνετ. Στο Μεξικό επίση αναφέρθηκε η σημασία τη απόφαση για την Νότιο Αμερική. οπότε ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση για όλο τον κόσμο. βέβαια, ε, ε, πολύ συχνά ε, σε τέτοιου περιπτώσεις το Συμβούλιο ε, για αντιδρώντας σκέφτεται να υποβάλει προσφυγή, έφεση εναντί του δικαστή της απόφασης αυτής και ενδεχομένως αυτό θα οδηγούσε σε περαιτέρω τροποποίηση των κανόνων πρόσβαση και διεύρυνση των εξαιρέσεων. Αυτό θα ήταν πολύ αρνητικό. Τρει μέρε μετά την απόφαση του δικαστηρίου πήγα σε ένα πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη για να ε, συναντηθώ με ένα καθηγητή εκεί και μου είπε ότι ε, έλαβε οκτώ φορές στο τα ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο την είδηση της απόφασης του δικαστηρίου. Οτιδήποτε σημαίνει εδώ στις Βρυξέλλες έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Δύο ακόμα λεπτά, ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. συζητούμε τον 1049 και την αδιατύπωσή του. Ας έχουμε υπόψη μας το εξή. Ε, ο 1049 αυτή τη στιγμή δεν πληρεί τις, όλες τις προδιαγραφές ε, του, της σύμβασης του άρχους. Ε, ή τη σύμβαση ε, του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόβαση σε δημοσία έγγραφα. Για παράδειγμα, τον ορισμό του εγγράφου, ε, η εφαρμογή τη δοκιμή του δημοσίου συμφέροντο στι εξαιρέσει, αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί. Ε, ακούσαμε, το, το ζήτημα, ακούσαμε τα σχόλια για το θέμα των γεωρικών επιδοτήσεων, πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε τα συμφέροντα, τα κρατικά με τα ατομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ε, υπάρχει ε, η, η επανάσταση των ανοιχτών δεδομένων ε, μέσω της, ε, είναι μια πρωτοβουλία μέσω της ε, οποίας τα κράτη-μέλη δημοσιοποιούν μεγάλα, μεγάλο αριθμό εγγράφων στο κοινό. Ε, ε, ε, για παράδειγμα κρατικές ενισχύσεις ε, αν γίνουν τροποποίησεις το 1049 θα πρέπει αυτές να οδηγούν προς την ευθυγράμμιση του με τις ελάχιστες προδιαγραφές ο περιορισμός της ε, κάλυψης είναι κάτι που δυσαρεστεί πολλούς. Θα πρέπει να ε, ε, διασφαλίσουμε επίσης ότι θα λειτουργεί στην πράξη ο κανονισμός ακόμα και να μην τροποποιηθεί. Ε, ο πρόεδρος λέει ότι πρέπει να τελειώνει ο ομιλήτρια. Πιο αργά και πρέπει να τελειώσετε κιόλα. Οπότε αυτά τα δύο πώ θα τα συμβιβάσετε δεν ξέρω. Ναι, πρέπει, πρέπει, πρέπει ακριβώ και εγώ να ισορροπήσω ανάμεσα στα δύο. Ε, ναι, θα κλείσω εδώ. Να πω το εξή. Ε, το και μόνο γεγονό ότι η σημερινή ακρόαση παρόλο να μην λάβει χώρα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Είναι πολύ σημαντικό ε, ε, άνθρωποι όπως εμείς εδώ πέρα να μπορούμε να ερχόμαστε και να ακούγεται τη φωνή μας. Είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Ε, και αυτό δεν γίνεται να συμβεί αν δεν λαμβάνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Έλεν. Και εγώ θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην Όναλτ Μπράουερ που βοήθησε να γίνει αυτή η συνεδρίαση, όπως και άλλους. Αλλά όνα, δεν περιμέναμε η αρχή της μερικής ε, ε, πρόσβασης να οδηγούσε τελικά σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε νέα νομολογία και θα δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Προς μεγαλύτερο άνοιγμα πιστεύω. Προχωρούμε λοιπόν. Δίνω το λόγο στον Τσέσσαρη Ανεστίνη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, που ε, είναι ε, αστική καθήκοντα επικεφαλής τμήματος. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, είναι ε, ένα νέο θεσμικό όργανο το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, με ιδιαίτερη προβολή προς τα έξω και θα θέλαμε να υπάρχει διαφάνεια και μεγαλύτερη μάλιστα διαφάνεια και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Πείτε μας λοιπόν κύριε Ονεστίνη πώ έχουν τα πράγματα. Φαντάζομαι η υπηρεσία σα θα έχει θεσπίσει κανόνε για την πρόσβαση στα έγγραφα. Ο κύριο Ανεστίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και συμμετέχω στην ε, σημερινή μας ακρόαση. Και ευχαριστώ και τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο πριν από μένα και έθεσαν ξεκάθαρα ε, τις ε, γενικές γραμμές και το πλαίσιο ε, του θέματος που συζητάμε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι νέος οργανισμός, άρχισε να υπάρχει από τις αρχές του έτους και έχουμε αναλάβει δέσμευση να συμμορφωθούμε τον κανονισμό 1049 που εκφράζεται ε, στα άρθρα και στους κανονισμούς ε, που ε, διέπουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και τώρα ολοκληρώνουμε την υιοθέτηση των κανόνων εφαρμογής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες από τη δημιουργία της υπηρεσίας μας έχουμε τους δικούς μας κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιλαμβανόμαστε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές των εφαρμοστικών ε, κανονισμών τους οποίους τώρα υιοθετούμε. Το σημείο αφετηρία, όπως για κάθε εφαρμοστικό κανονισμό, είναι ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αφορά και μεμονωμένα άτομα και νομικά πρόσωπα καλύπτονται όλα τα έγγραφα ανεξάρτητα της, ε, του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα και ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού 1049 και βέβαια οι εξαιρέσεις του κανονισμού 1049. θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον κανονισμό και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού. Πάντω σε αυτά βασίζονται οι εφαρμοστικές διατάξεις Εάν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση λάβει ένα αίτημα για έγγραφα από κάποιο τρίτο φορέα, και αυτό για τη δική μα περίπτωση είναι σημαντικό, γιατί τα περισσότερα έγγραφα τα οποία έχουμε ε, πολύ συχνά προέρχονται από τρίτους ε, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποφασίζουμε ποιες εξαιρέσεις ισχύουν και τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τα έγγραφα. Και θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το έργο. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, θα ορίσει ένα συντονιστή πρόσβαση στα έγγραφα μέσα στην υπηρεσία μας. Ε, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με κάποιες από τις συστάσεις που ακούσαμε νωρίτερα από προηγούμενους ομιλητές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζεται πλήρως ο κανονισμό στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ότι θα χειριζόμαστε τα αιτήματα σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον κανονισμό. Θεσπίζουμε κάποιες νέες διαδικασίες και θεωρώ ότι ο σημαντικός ρόλος του συντονιστού της πρόσβασης στα έγγραφα θα διασφαλίζει και την σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση. Αυτή η σωστή πληροφόρηση θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που προέρχεται από διάφορα θεσμικά όργανα και προέρχεται και από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβαδίζει με αυτά που ανέφερε ο διαμεσολαβητής προηγουμένως. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ε, μια κοινή κουλτούρα και μια κοινή κατανόηση του κανονισμού. Γι' αυτό θέλουμε μέσα στην υπηρεσία μας να έχουμε σωστή κατάρτιση για όλους τους υπαλλήλους, ούτως ώστε να έχουμε κοινή αντιμετώπιση και όλοι να κατανοούμε κατά τον ίδιο τρόπο το πώς εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις. Επαναλαμβάνω, επειδή προέρχονται από διαφορετικέ υπηρεσίε και από διαφορετικέ χώρε, όταν έρχονται στην υπηρεσία μα θα φροντίζουμε με τη σωστή κατάρτιση να διασφαλίζουμε ότι όλοι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Αυτοί οι εφαρμοστικοί κανόνε, του οποίου τώρα θεσπίζουμε, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, ελπίζουμε, αρκετά σύντομα. Θα πρέπει πρώτα να οργανωθεί η υπηρεσία μα, και βλέπετε ότι ε, αυτή ότι οι κανονισμοί είχαν προτεραιότητα για την υπηρεσία μας και γι' αυτό ήδη ασχολούμεθα με τη θέσπιση αυτών των εφαρμοστικών διατάξεων. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Ονεστίνη. Έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι από το Συμβούλιο που πάντα ήταν πιο διστακτικό όσον αφορά το να μοιράζεται περισσότερα στοιχεία εξωτερικών σχέσεων με τις πολίτες η Φωτή και Διαμαντούρο. Θαυμάζω τη διπλωματική σας προσέγγιση, της δεξιο, επιδεξιότητάς στη διπλωματική κυρία μου. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Τον Χιούμπερτ Σασλεύσκη καλό τώρα, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με θέματα καλύτερης διοικητικής πολιτικής και κανόνων να εξηγήσει αυτό πώς είναι η προϋπόθεση ε, η διαφάνεια για μια ανοιχτή και πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Κύριο Σλασεύσκη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους εισηγητές για αυτή την πρόσκληση που μου απευθύνθηκε, που ήρθε έγκαιρα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα που είμαι σχετικά νέος στον τομέα αυτό. Ακούγοντας κάποιες από τις παρεμβάσεις, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια πολιτική των θεσμικών οργάνων για το, ε, να μπλοκάρει την πρόσβαση των ε, πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και όπως είπε ο ε, Μπάνιον, οι δεινόσαυροι φυλάνε αυτά τα μαύρα μυστικά και δεν αφήνουν να βγουν στο φως. Προβάλλονται συνήθως ακραίες περιπτώσεις όταν συζητάει κανείς ε, εν είδη επιχειρήματος. Μιλώ εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είστε βέβαιοι ότι η κατάσταση δεν είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται. Και εγώ δεν αισθάνομαι σαν τυρανόσαυρου Ρέξ. Ε, η κατάσταση είναι πολύ πιο θετική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τα όσα είπε η κυρία Γιάτεν Μάκη. Δηλαδή είναι σημαντική διαφάνεια εξασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, προωθεί την ορθή διακυβέρνηση και αυτές είναι έννοιες τις οποίες υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να είναι ανεξαρτητή, ανοιχτή και διαφανής ε, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω της κοινοτικής μεθόδου και την υπερασπιστήκαμε αυτή τη μέθοδο, την ανοιχτή και την ε, ε, ολιστική της διακυβέρνησης. Πώς το εφαρμόζουμε στην πράξη. Ξεκινήσαμε αρχή της δεκαετίας του 90. Έκτοτε έχουν αναλυφθεί διάφορες πρωτοβουλίες. Η πιο σημαντική είναι ο κανονισμός 1049. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεκάλυψε πολλά έγγραφα, διέθεσε πολλά έγγραφα αυτοβούλους και δυνάμει του 1049. Κάποια στοιχεία να παραθέσω. Για τα αιτήματα που υπευλήθησαν στα πλαίσια του 1049 και ποια έγγραφα χορηγήθηκαν. Τα αιτήματα, τα αιτήματα, όχι αριθμό εγγράφων. 2001. Περίπου 500 αιτήσει λάβαμε. Πέρσι πάνω από 6.000 πάνω από 80% από αυτά τα έγγραφα χορηγήθηκαν. Και περίπου 150 ε, τα εξετάζει, εξετάζει τη χορήγησή τους ο Γενικός Γραμματέας μετά από έφεση αν θέλετε. Άρα το σύστημα λειτουργεί. Κάποιοι ομιλητές αναφέρθηκαν στις καθυστερήσεις και ε, αμφισβήτησαν κάποιες αποφάσεις όταν οι αποφάσεις ήταν αρνητικές. Η κυρία Μπερτιέ είπε ότι ζητείται παράταση χρονική ακόμα και αν κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται. Σας διαβεβαιώ, όταν ζητείτε χρονική παράταση υπάρχει πάντα ένας σοβαρός λόγος για κάτι τέτοιο. Διότι και εμείς Πιστεύουμε ότι όσο πιο γρήγορη η ανταπόκριση, τόσο, και, τόσο πιο αποδοτική θα είναι. Πολλές αιτήσει όμως είναι περιπλοκότατες. Χρειάζονται έρευνα. Και παρόλο που ο κύριος Διαμαντούρος είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε αρκετό προσωπικό για να ανταποκρινόμεθα, ποτέ δεν θα έχουμε αρκετό προσωπικό. Και στην παρούσα κατάσταση είναι απίθανο να υπάρξει βελτίωση. Δεν θα δικαιολογηθώ μέσω της ελλείψεως πόρων. Αυτό είναι ένα μικρό στοιχείο, αλλά σημαντικό. Κάτι πιο σημαντικό. Οι αιτήσει όπως τα βλέπει ο υποβάλλον την αίτηση, όπως βλέπει την αίτηση αυτός που την υποβάλλει, δεν βλέπει ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που θα πρέπει να σταθμιστούν όταν υποβάλει κάποιο αίτηση. Τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρει πίν και πρέπει να διαφυλαχθούν κάποια πραγματικά σημαντικά συμφέροντα. Και είναι στο σταυροδρόμι όλων των συμφερόντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να σταθμίσουμε σωστά τα συμφέροντα. Διαφορετικά θα χάσουμε την υπόθεση στο δικαστήριο και δεν χάνουμε την υπόθεση στο δικαστήριο, διότι δεν ανοίγουμε ένα χαρτοφυλάκιο ή χορηγούμε ένα έγγραφο, καμιά φορά χάνουμε γιατί έχουμε δώσει το έγγραφο. Άρα χρειάζεται μια καλή ισορροπία. Και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι θα επιθυμούσαμε. Έχω αναλάβει το θέμα της διαφανείας εδώ και δύο εβδομάδες. Θα κάνω ότι μπορώ να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Διότι δεν λειτουργεί έτσι μια καλή διοίκηση. Ταυτόχρονα όμως σας ζητώ να καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Τώρα η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Αυτό είναι ένα στοιχείο της διαφάνειας. Υπάρχουν και άλλες στοιχείες όμως της διαφάνειας. Και θα ήθελα να τις αναφέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρότεινε την νομοθεσία και προτείνει νομοθεσία πολύ συχνά έρχεται σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών η διαμόρφωση πολιτική μέσω δημόσια διαβούλευση και διασκέψεων στι οποίε συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα μέρη και έχουμε θέσει κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ για τη διαβούλευση με του εμπλεκομένου φορεί και έτσι το κοινό πληροφορείται σωστά. Ε, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τι απόψει του. Έχουμε εξασφαλίσει και το ότι διατίθενται όλο και περισσότερες πληροφορίες μέσω δημοσίων αρχείων και οι προτάσεις του συναδέλφου του Γραφείου Δημοσιεύσεων είναι και αυτές στοιχεία για την βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα. Καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν θα επισέθω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, θα ήθελα να πω ότι δεν ενημερώνονται διάφοροι φορείς, ότι οι διάφορες υπηρεσίες ότι λόγω της, ε, της ε, συνθήκης της Ζαβώνας θα πρέπει να συμμορφωθούν και αυτές με τους νέους κανόνες. Σας λέω και Διαμαντούρο ότι θα κάνουμε τα δέοντα για να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το τι πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Λασεύσκη. Έχουμε 10 λεπτά για συζήτηση. Θα ήθελα να καλέσω τον διαμεσολαβητή να λάβει το λόγο βέβαια ε, πρώτα, αλλά μετά θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κ. Διαμαντούρος. Ε, σημείωσα τα όσα είπε η κυρία Ντάρμπισερ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η καινούργια νομολογία. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτή. Να κάνω δύο-τρία σχόλια συνοπτικά για, τα, για του κ. Σλαζεύσκη. Καταρχήν να σας συγχαρώ που αναλάβατε τα καθήκοντά σας πολύ πρόσφατα. Δύο εβδομάδες αν κατάλαβα καλά έχετε σε αυτή τη θέση. Ωραία, σας εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία. Να σας πω δύο-τρία πράγματα, αν μου επιτρέπετε, όχι ως διαμεσολαβητής, εξωτερικός δηλαδή μηχανισμός ελέγχου, αλλά ως διαμεσολαβητής που είναι σημαντική πηγή πληροφοριών για τα θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένη και τη δική σα διεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι η Κομισιόν σε πολύ ψηλό επίπεδο είναι προσιλωμένη στη διαφάνεια και είναι αλήθεια ότι σε πολύ ψηλό επίπεδο το εκφράζει ε, πολύ δραστήρια. Το πρόβλημα είναι όταν κατεβαίνει κανεί στα χαμηλότερα κλιμάκια. Το πρόβλημα είναι το πώς αυτή η δέσμευση των υψηλών κλιμακίων της κορυφής εφαρμόζεται στην πράξη από τον Α ή το Β υπάλληλο, ο οποίος ε, ε προσπαθεί να καλύψει τα νότα του. Συνεπώς δεν αμφισβητώ την θεσμική δέσμευση και προσήλωση της Κομισιόν σε υψηλό επίπεδο. Ο Γενικός ε, Γραμματέας πάντοτε μας υποστηρίζει. Το θέμα είναι το πώς εκπαιδεύετε τους συναδέλφους σας στην εφαρμογή όλων αυτών. Γιατί η εφαρμογή απαιτεί μια λήψη απόφασης κάθε φορά και είναι προσωπική ευχέρεια η απόφαση. Συνεπώς ε, ε, χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού. Η Επίτροπος ο, μάλλον ο Επίτροπος σχολίασε μια παλιότερη ε, ε, περίπτωση ε, για μια, ε, ασχολήσει με παλιότερη επίφωση, ε, απο, απόφαση της Κομισιόν η οποία είχε ζητήσει 15 φορές παράταση και χρειάστηκε να παρέμβω εγώ για να δοθεί μια απάντηση. Με, τις περισσότερες φορές υπάρχουν σοβαροί λόγοι της παράτασης, αλλά όχι πάντοτε. Τέλος. Για το θέμα του, της του προσωπικού. Το καταλαβαίνω. Πραγματικά το καταλαβαίνω, το κατανοώ μπορώ να πω. Από τη δική μου οπτική γωνία, ως διαμεσολαβητή δηλαδή, ε, το επιχείρημα της έλλειψης προσωπικού δεν είναι επαρκέ, ιδιαίτερα ενώ σε ό,τι αφορά τον πολίτη. Εγώ δεν μπορώ να πω ω διαμεσολαβητή, έτσι. Δεν μπορώ να επικαλεστώ ε, έλλειψη προσωπικού. Έλλειψη προσωπικού σημαίνει κακή διοίκηση. Πρέπει να βρείτε μια λύση. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό στον πολίτη. Δεν μπορώ να του πω δεν έχουν αρκετό προσωπικό, το προσωπικό είναι διακοπέ. Καταλαβαίνετε έτσι. Ε, δύο ακόμα σχόλια. Ίσως δεν κατάλαβα πολύ καλά το τι είπατε και ζητώ συγγνώμη αν έχω παρεξηγήσει. Αλλά αν πράγματι ισχύει πως η Κομισιόν λέει σκέφτεται να προσέξουμε μήπως και χάσουμε το δικαστήριο, δεν είναι σωστή. Το δικαστήριο αποφασίζει το πώς θα εφαρμόζει το 1049. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει νομική υπηρεσία στην Κομισιόν να σας συμβουλεύει σε περίπτωση που υπάρχουν έτσι παγίδες ή δυσκολίες. Και η νομική υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να σας προστατεύσει. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά είναι δική σας ευθύνη να είστε... Ε, ε να, να παίρνετε πρωτοβουλίες εκ των προτέρων. Ε, και βέβαια μη, έχω και εγώ το προσωπικό συμφέροντα, συμφέρον αν πηγαίνουμε συνεχώ στο δικαστήριο, κανένα δεν θα έρχεται στο διαμεσολαβητή, καταλαβαίνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ε, υπηρεσίε και τα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1η Ιουνίου θα συναντηθώ με όλου και έτσι κι αλλιώ σε κάθε χώρα που επισκέπτομαι, επισκέπτομαι και τι αντίστοιχε ευρωπαϊκέ ε, υπηρεσίε για να του ενημερώνω κι εγώ κι Ευχαριστώ πολύ. Μάικλ Κάσμαν και μετά η Ελένη. Ε, σπάνια υπερασπίζομαι άλλα θεσμικά όργανα. Όχι, όχι, λάθος και πάλι έκανα. Νομίζω ότι ε, είναι, ε, χρειάζεται και αυτό που και που. Χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερο προσωπικό, έτσι ώστε να φέρουμε πέρα στις δημοκρατικές μας υποχρεώσεις. Αλλά είναι τόσο αρνητική η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι πολιτικοί δεν θέλουν να εγκρίνουν περισσότερο προσωπικό στα θεσμικά όργανα για να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Συνεπώς είναι ένας φαύλος κύκλος και ε, αποτελεί τμήμα του προβλήματος. Η, η πολιτική μας, οι γέτες σε όλα τα όργανα ε, θέλουν να προστατεύσουν τα νότα τους και το γνωρίζουν όλοι αυτό. Οπότε αυτό που είναι αναγκαίο είναι μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική νοοτροπία. Έτσι ώστε οι επικεφαλής όλων των οργάνων να ε, καταλάβουν ότι πρέπει να απαιτήσουν περισσότερο προσωπικό προκειμένου να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους που απαιτείται ε, κάτι που απαιτείται από την κοινωνία των πολιτών, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Γιατί αλλιώς αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι πολίτες. Η Χέλεν. μια πρόταση προς τον κύριο Σαζεύσκη, μια και μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, είναι φρέσκος. Ε, να μην ε, σκέφτεστε το σύστημα πρόσβαση των εγγράφων μόνο από, από μέσα, αλλά και απ' έξω. Να σκέφτεστε τι χρειάζεται να ξέρει ο πολίτης προκειμένου να ζητήσει έγγραφα και να έχει πρόσβαση. Είναι πολύ καλό ότι αυξήθηκαν αιτήσει από 5 σε 6.000, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρό το νούμερο σε μια περιοχή 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Πολύ δε περισσότερο που γνωρίζω ότι οι περισσότερε αιτήσει προέρχονται από ε, ε, ελάχιστε ε, μη κυβερνητικέ που έχουν έδρα τι Βρυξέλλες. Ε, εγώ ρώτησα, έχω ρωτήσει με κυβερνητικέ οργανώσει σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αν ξέρουν πώ να υποβάλουν αίτημα και πολύ συχνά δεν ξέρουν και δεν μπορούν. Μπερδεύονται. Μετά. Ε, και ακόμα και όταν μας δίνονται πληροφορίες αυτές είναι στα αγγλικά ή γαλλικά Σχεδόν ε, κανένα ε, site της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, έχει πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορεί κανείς να υποβάλει έτοιμα. Η Γενική Γραμματεία ίσως να είναι ε, ένα site. Οπότε οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν την, τη Γενική Γραμματεία, ξέρουν την τάδε Γενική Διεύθυνση, την τάδε ε, υπηρεσία ή οργανισμό κλπ. Και πάνε εκεί και βλέπουν ότι δεν έχει τίποτα στη γλώσσα του. Οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί περισσότερο ο κόσμο για το πώ μπορεί να κάνει αιτήματα για πρόσβαση έγγραφα. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ, λέει πρόεδρο, μία ερώτηση στον κύριο Σλαζεύσκη και δεν ξέρω πώ θέλει και κανεί άλλο να σχολιάσει. Νομίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο την ανάγκη και το ίδιο το κοινοβούλιο να γνωρίζει, όχι μόνο οι πολίτες βέβαια, τις, ε, τις ε, βάσεις πάνω στις οποίες διαπραγματεύεται η Κομισιόν Διεθνής Συμφωνίες. Όπως γνωρίζετε κύριε Σλαζεύσκη, έχουμε, έχουν διεξαχθεί πολλές διαθεσμικές και συγκρούσει ανάμεσα στο Συμβούλιο και τα άλλα όργανα, έτσι ώστε να, το Κοινοβούλιο να γνωρίζει τι διαπραγματευτικέ εντολέ που χρησιμοποιούν ε, οι ε, υπηρεσίε Κομισιόν όταν διαπραγματεύονται ε, ε, τις ε, θέματα, σε, θέματα εσωτερικών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. πιστεύετε ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί η πρόσβαση των πολιτών και σε αυτά τα έγγραφα, διότι και αυτά τα έγγραφα ε, επηρεάζουν πάρα πολύ άμεσα την καθημερινή του ζωή και τα δικαιώματά τους. Ο κ. Λαζεύσκη. Να απαντήσω σε όλα όσα σχολιάστηκαν. Καταρχήν ε, για το θέμα του προσωπικού. Ε, είναι ένα θέμα που επανέρχεται, της Αρεφρέν. Συμφωνώ με τον κύριο Διαμαντούρο δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού ως δικαιολογία. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός. Και είναι ένα γεγονός, ένα εμπόδιο αξεπέραστο, ανυπέρβλητο πολλές φορές. Οπότε ε, είναι σαν να έχει ε, δύο λεπτά και να έχει πολλά να πει όπω η κυρία Ντέρμπισάιρ <laughs> προηγουμένως. Ε, Μερικέ φορέ είναι αδύνατον, είναι, βρισκόμαστε σε, σε, πολύ δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω βέβαια. Αυτό είμαι υπεύθυνο και για τι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό και για διάφορα θέματα εσωτερικού έλεγχου της Κομισιόν. Ποτέ δεν έχουμε δεχτεί τη δικαιολογία ότι δεν είχαμε αρκετό προσωπικό γι' αυτό δεν το κάναμε. Όμω, η κατάσταση σημαίνει ότι από κάπου πρέπει να κόψουμε και κόβοντας και κόβοντας και περικόπτοντας φτάνει σε ένα σημείο που ε, περικόπτεις και σημαντικές δραστηριότητες. Δεν πάση περιπτώσει, εκτός θέματος βέβαια αυτό. Ε, λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου το σχόλιο ότι πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα από την πλευρά και από τη σκοπιά του πολίτη. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε πράγματι. πρωτοβουλίες όπως αυτή του υπηρεσία δημοσίευσεων ε, έχουν ως ε, στόχο να γίνει πιο ε, σαφές ε, το σημείο εισόδου για, ένα, για μια μεγάλη κατηγορία πληροφοριών. Να μην χρειάζεται κανείς να μπει στο Europa, να μπορεί να βρει αυτά τα έγγραφα πολύ πιο εύκολα και αυτές τις πληροφορίες. Η δυσκολία είναι ότι υπάρχει τόσος μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο, κατοντάδες χιλιάδες σελίδων, που και αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονό ότι θέλει κανεί να είναι πιο ανοιχτό. Αλλά όσο πιο πολλέ είναι οι πληροφορίε, τόσο πιο δύσκολο είναι να αναζητήσει και να βρει κάποιο την πληροφορία που τον ενδιαφέρει σε αυτόν τον όγκο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε βέβαια την κατάσταση. Εγώ πολύ συχνά αυτό που κάνω όταν χάνομαι είναι βάζω τη, τη, ε, λέξη κλειδιά στο Google και βρίσκω τα έγγραφα που χρειάζομαι τελικά. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τι γλώσσε, είναι θέμα ε, προπολογισμού, είναι θέμα οικονομικό. Προσπαθούμε να έχουμε προτεραιότητες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά το πιο σημαντικό, μάλλον πιο δύσκολο ερώτημα ε, που ετέθη στο τέλος από την πρόεδρο, του κ. Χαουτάλα, ε, είναι ότι η απάντηση βρίσκεται στην ε, διοργανική συμφωνία. Η διοργανική συμφωνία, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ε, ε, μπορεί να ρυθμίσει το θέμα και δεν θα ήθελα να σχολιάσω εγώ. Κύριε Χαουτάλα, τα δικαίωμα των πολιτών ενδεχομένως ε, θα πρέπει να διευρυνθεί και στα άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων. Ε, ενδεχομένως λέω γιατί ο πολίτης ανήκει και σε μια παγκόσμια κοινότητα Οπότε θέλει να ξέρει τι κάνουν οι εκπρόσωποι του εξ ονόματός τους στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες για θέματα ποιότητας τροφίμων, ε, και ίσως να υπάρχει και εκεί ένα θέμα προστα... Ε, ε, ευθύνης προστασίας, αλλά θα ήθελα να το θέσω και στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει σκέψη, ναι. Όπως είπα και στην αρχή όμως ε, βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας καθορισμού των εσωτερικών κανόνων. Τώρα ξεκινάμε και προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τις αντικρώμενες ανάγκες. Ε, θα πρέπει να κάνουμε μια διακρισία ανάμεσα στον 1049, το είπα και πριν αυτό, που αφορά όλους τους πολίτες και την πρόσβαση που θα πρέπει να έχουν οι ευρωβουλευτές η ανώτατη εκπρόσωπό μα ε, το σχολίασε σε συζητήσει με το Κοινοβούλιο και σε δηλώσεις για την πολιτική λογοδοσία. Στην, ε, έχει επιβεβαιώσει δηλαδή ότι ακόμα και σε αυτή την μεταβατική φάση δεν ε, θα περιορίσουμε τα γεκτημένα. Θα πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση χωριστά για να διαπιστώσουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν κενά. Υπάρχει μια καλή θέληση ε, μια καλή πρόθεση εκ μέρους της Κομισιόν. Τώρα κάποια από τα θέματα σχετίζονται και με τις ε, συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα ήδη ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις ε, διαοργανικές ε, συμφωνίες συγκεκριμένα. Δεν είμαι ειδικό σε αυτό, αλλά ε, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας ακόμα και αν πολλά από τα έγγραφα τα οποία χειριζόμαστε ε, θα υπάρχουν τους κανόνες ε, των διοργανικών συμφωνιών, γίνονται συζητήσεις ε, και υπάρχει και η πολιτική βούληση που έχει εκφράσει η υπατή εκπρόσωπος αντιπρόεδρος Κομισιόν. Ωραία. Θα δώσω το, την προεδρία στον Μάικλ αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ. Thank you Κάσμαν, ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω από τους, κυρίου, τους επόμενους ομιλητές να έρθουν στο βήμα. Κέρτιν, Χάστινγκς, Βαλέριο Πλάκο και Παναρέλα.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 με τίτλο «Προκλήσεις για την αναδιατύπωση ή αντικατάσταση του κανονισμού 1049 του 2001 στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας». Όσο ενδιαφέρουσες και αν είναι οι συζητήσεις ε, μεταξύ σας, θα σας παρακαλούσα να κάνουμε ησυχία για να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι ομιλητές από το βήμα. Ξεκινάμε με κάποιον που ήδη γνωρίζετε από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, την καθηγήτρια Ντέιδρα Κέρτιν, που είναι και υπεύθυνη για το ε, τμήμα ε, δικαίου και διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, καθώ και στο Πανεπιστήμιο τη Ουτρέχτη. Το 2007 της απονεμήθηκε το βραβείο Σπινόζα από την ε, Ολλανδική Ένωση Επιστημόνων για την έρευνά της στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης και πρώτη φορά δόθηκε αυτό το βραβείο Σπινόζα σε νομικό. Το 2008 τη δόθηκε από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου ε, το, ο επίτιμος τίτλος του διδάκτορος. Κύριε κυρία Ντέιντε Κέρτιν έχει το λόγο και θα προσπαθήσω κι εγώ όπως οι προηγούμενοι πρόεδρος ε, να είμαι αμήλικτος στο χρόνο που σας διαθέτω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Περνώ κατευθείαν στο θέμα, αφού δεν έχω πολύ χρόνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα το πρωί να μιλήσω σε αυτή την ακρόαση. Ως ακαδημαϊκός, εγώ θα ήθελα να δω τις προτινόμενες αλλαγές στον κανονισμό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας που έχει τεράστια σημασία για τον τομέα αυτό. Στην οθόνη μπορείτε να δείτε τα, τις βασικές γραμμές αυτών που θα αναφέρω στην παρουσίασή μου. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καταρχήν διότι όπως ακούσαμε διευρύνει το πεδίο εφαρμογή. Δεν μιλάμε μόνο για τα τρία θεσμικά όργανα αλλά για όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ανεξάρτητα με το πότε και αν τροποποιηθεί ο κανονισμός, δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνθήκη της Λισαβόνας είναι διότι η ανοιχτή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων βασίζεται στο άρθρο 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επανέλθω σε αυτό εντό ολίγου. Και τρίτος λόγο, για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνθήκη τη Λισαβόνα σε αυτό το πλαίσιο είναι η έμφαση που δίδει στην δημοκρατία και στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην έννοια της ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Πρώτη φορά μπαίνει στην συνθήκη κάτι τέτοιο, διατυπώνεται στο άρθρο 10 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τις παραμέτρους ε, του αν ε, πριν από 10 χρόνια εγκρίθηκε ένας κανονισμός. Είναι διαφορετικό το νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή και αυτό θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτά που είναι στην οθόνη, ούτε εγώ μπορώ καν να τα διαβάσω. Προσπάθησα να έχω ε, λίγε διαφάνειε γιατί δεν είχα χρόνο. Δυστυχώ δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε πολύ καλά. Το πρώτο σημείο είναι ότι η ανοιχτή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων και η αρχή του ανοιχτού χαρακτήρα είναι κάτι το οποίο ε, τονίζεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και πρόσβαση στα έγγραφα και συμμετοχή των πολιτών. Είναι δύο πτυχές που ε, διασυνδέονται και διατυπώνεται στη συνθήκη ως συγκεκριμένο πολιτικό δικαίωμα. Είναι μια δημοκρατική αρχή το οποίο τονίζεται στο άρθρο 10 και αυτό αποτελεί πλέον τον ε, χρυσό κανόνα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τον κανονισμό για την πρόσβαση σε έγγραφα και δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε αυτόν τον κανονισμό για να διασφαλίσουμε την ε, διαφάνεια. Θα πρέπει να το δούμε μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε η εκτελεστική εξουσία, είχε το Συμβούλιο των Υπουργών που ήταν η νομοθετική εξουσία επί πολλά έτη και υιοθετούσε την νομοθετική, το νομοθετικό του έργο ε, ε, αλλά τώρα έχει αλλάξει το μοντέλο και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, ιδίως με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας σαφώς τονίζει αυτή την αλλαγή μοντέλου και γι' αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι το δικαστήριο σε πρόσφατες αποφάσεις του για την πρόσβαση στα έγγραφα λέει προς το Συμβούλιο ότι έχετε μπει στην νομοθετική διαδικασία και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναφέρονται τα ονόματα μεμονωμένων κρατών μελών. Μπορούν να αναφέρονται ποια ήταν τα κράτη-μέλη αυτή είναι η τωρινή κατάσταση. Στην απόφαση Τούρκο που αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, τόνισε το δικαστήριο πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια στην νομοθεσία. Από την υπόθεση Τούρκο και μετά, αυτό το οποίο εγώ παρατήρησα είναι ότι ορισμένα θεσμικά όργανα έχουν την τάση να λένε ότι καλός όσον αφορά τη διαφάνεια, αλλά εδώ απαιτείται λιγότερη διαφάνεια για τα διοικητικά θέματα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όμως σε αυτό το σημείο, διότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ο κανονισμός για την πρόσβαση στα έγγραφα είναι ακριβώς για να διασφαλίσει ότι η διοίκηση θα είναι διαφανής αν σκεφτούμε την δημοκρατία στα θέματα διοίκηση και στα κράτη-μέλη, ακριβώ για αυτού του λόγου και για λόγου λογοδοσία ε, υπάρχει αυτό ο κανονισμό. Υπάρχει μια υπόθεση σε κρεμότητα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με αεροπορικέ μεταφορές όπου και πάλι για λόγους ε, λογοδοσίας ε, και ε, διαφάνειας τονίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό οι πολίτε να γνωρίζουν τους λόγους. Ξεκίνησα από τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία τονίζει ιδιαίτερα την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας θα πρέπει να δούμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν μιλώ για δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο υπάρχει και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο πράγμα όπως στα κράτη-μέλη. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια που αποτελούν πυλώνες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ε, καταργήσει την κυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, θα χρειαζόμασταν μεγαλύτερο βαθμό ε, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. και η ανοιχτή προσέγγιση δεν υποκαθιστά το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και δεν πρέπει να νοείται ως εναλλακτική λύση προς αυτό. Είναι απλώς κάτι το οποίο ενισχύει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι η ανοιχτή προσέγγιση καλύπτει και τα νομοθετικά και τα διοικητικά θέματα. Η πρόσβαση σε έγγραφα πρέπει να νοείται όχι ως ένα προσωπικό δικαίωμα, όχι ως κάτι το οποίο ε, οφείλει η διοίκηση ως διαδικασία, πρέπει να νοείται ως συλλογικό θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες, χωρίς να χρειάζεται καμία ιδιαίτερη αιτιολογία. Είναι τμήμα της δημοκρατικής κληρονομιάς των πολιτών. Τρία λεπτά έχουν μείνει ακόμη για την ομιλήτρια. Έχω άλλα δύο σημεία να τονίσω. Ένα από αυτά τα σημεία αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε την ανοιχτή προσέγγιση. Λέγεται πολλές φορές ότι οι εξωτερικές σχέσεις εξαιρούνται γιατί είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας ή εξωτερικών σχέσεων και εξαιρούνται. Επανερχόμενοι στις βασικές αρχές, στο άρθρο 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να πω ότι όλος ο τομέας των εξωτερικών σχέσεων και η ΚΕΠΑ και αυτό το οποίο αποκαλούσαμε κοινοτική αρμοδιότητα στα θέματα των εξωτερικών σχέσεων καλύπτονται από την έννοια της ανοιχτής προσέγγισης. Το αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών περιλαμβάνει διατάξεις που είναι δεσμευτικές για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα παράδειγμα είναι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα που αποδεικνύει αυτό το οποίο θέλω να σας πω. Πρέπει να δούμε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε εξαιρέσεις. Όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού, αυτό το οποίο μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι χρειάζεται η εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος στην δημοσίευση εγγράφων και του δικαιώματος διαφύλαξης του απορρίτου. Ένα σημείο το οποίο αναφέρθηκε εν συντομία σήμερα το πρωί είναι το θέμα ε, της διαβάθμισης εγγράφων και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί ακόμη επαρκώς. Ξεκινώντας από την κληρονομιά του παρελθόντος, πολλά θεσμικά όργανα ε, θεωρούσαν ότι μπορούν από μόνο τους να αποφασίζουν τι θα αποκαλύπτουν και τι όχι. Πρέπει πλέον να υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς ε, και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ίδιο επίπεδο ε, όπως και η διοικητική πρόσβαση στα έγγραφα. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια σοβαρή, ανοιχτή συζήτηση στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το όλο σύστημα καθορισμού του απορρίτου δεν θα υπονομεύει τις διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφα και την ανοιχτή προσέγγιση. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω κάτι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας βοήθησε πάρα πολύ να θέσουμε τις γενικές αρχές, αλλά το Δικαστήριο μπορεί μόνο κατά περίπτωση να εξετάζει τις διάφορες ε, αποφάσεις τις οποίες ε, εκδικάζει. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους νομοθέτες και την ανοιχτή δημόσια συζήτηση. Επί τη βάση των αρχών που ήδη υπάρχουν τώρα και στη συνθήκη της Λισαβόνας και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα πρέπει οι νομοθέτες και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά και η Επιτροπή στην προπαρασκευαστική φάση, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Professor. Ευχαριστώ καθηγητά Κέρτιν. Θα κάνουμε σύντομη παρουσίαση κάποιου που είναι γνωστό σε όλους στο Κοινοβούλιο. Του Πίτερ Χάστινγκς, του Ευρωπαϊκού Ποπτήρου, προστασία των δεδομένων. Είναι σε αυτή τη θέση από τον Ιανουάριο του 2004 και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι ε, ο Ευρωπαίος για την υποπτία των δεδομένων είναι ένας του συνήθις υπόπτους που είναι εδώ, που συζήτησε τον κανισμό για την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα και χαίρομαι και αυτό διότι επιβεβαιώνεται έτσι ότι η προστασία των δεδομένων και η διαφάνεια των κυβερνήσεων είναι αλληλένδετα. Η διαφάνεια, η ιδιωτική ζωή, η προστασία των δεδομένων είναι μεταξύ ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα της χάρτας και αντικατοπτρίζονται και στη συνθήκη όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι δίπλα-δίπλα σαν διατάξεις γενικής εφαρμογής. Εξυπακούεται ότι η σημασία που έχουν αυτά τα δικαιώματα για την κοινωνία αυξάνεται συνεχώς λόγω της εντυπωσιακή επέκτασης της κοινωνίας των πληροφοριών όπως αποκαλείται και σε αυτό το πλαίσιο ο καθορισμός, ο αυτοκαθορισμός της διαθέσεως των πληροφοριών ξεπερνά ε, τα όρια του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων συγκεκριμένου ατόμου και σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων ε, για, που επηρεάζουν τη ζωή του. Αυτό συνεπάγεται διαφάνεια του ιδιωτικού τομέα καθώς και διαφάνεια των κυβερνήσεων. Όσον αφορά τις κυβερνήσεις, οι πολίτες έχουν δικαίωμα και στα δύο να υπάρχει ανοιχτή και ελεγχόμενη κυβέρνηση και μια κυβέρνηση που εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ε, τα επεξεργάζονται με νόμιμο και δίκιο τρόπο. Καμιά φορά η διαπάνη προστασία των δεδομένων, η προστασία τη προσωπική ζωή, ίσω να οδηγεί σε αντίθετε διεκδικήσει. Κανονικά ταιριάζουν και ενισχύουν η μία πτυχή την άλλη και έτσι τελικά ε, αποκτά την εμπιστοσύνη του λαού κυβέρνηση. Να πω ξανά, ότι ο ρόλος προστασία των δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή, δεν είναι η παρεμπόδιση της προσβάσεως του κοινού στις πληροφορίες όταν αυτό συνεπάγεται σε προσωπικά δεδομένα. Για να εφαρμόζονται οι κανόνες πρέπει να εφαρ... Εάν εφαρμοστούν έτσι οι κανόνες για ιδιωτική ζωή, θα μειωθεί η διαφάνεια της ευρωπαϊκής διοίκησης, αλλά και θα υπονομεύεται και η αξιοπιστία της προστασίας των δεδομένων, αυτής καθ' Η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους υπάρχει πρόσβαση του κοινού στα προσωπικά στοιχεία και μπορεί να θεωρηθεί αυτή ως νόμιμη. Προφανώς υπάρχουν πολλές προσωπικές ε, πληροφορίε που η αποκάλυψη αυτών δημοσία δεν θα ήταν νόμιμη χωρίς σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Προφανέ παράδειγμα ιατρικά ε, δεδομένα για το προσωπικό κλπ. Α, όμως, κάποιες γενικές πληροφορίες, ή καθαρά επαγγελματικές πληροφορίες μπορούν να δημοσιευθούν και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από τη στιγμή που εξασφαλίζεται ότι προστατεύονται τα νόμιμα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Φτάνουμε στην περίφημη περίπτωση της Bavarian Lager στο δικαστήριο όπου σβηνόταν τα ονόματα των εκπροσώπων των επιχειρήσεων από τα πρακτικά των συνεδρίων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφαση του περσινού Ιουνίου, το Δικαστήριο συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αποκάλυψη των πέντε ονομάτων δεν θα τέριαζε με του κανόνε τη προστασία των δεδομένων. Αυτή ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμω, το συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε από αυτή την υπόθεση δεν θα πρέπει να είναι ότι αυτέ οι πληροφορίε μπορούν μόνο να διατίθενται δημόσια εάν ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί. Κατά την άποψή μου το συμπέρασμα θα έπρεπε να είναι το εξή. Η δημόσια αποκάλυψη θα μπορούσε να τέριαζε με τους κανόνες για προστασία των δεδομένων αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δράσει διαφορετικά πριν τη στιγμή που δημοσιοποίησε αυτά τα ονόματα. Η αποκάλυψη των πέντε ονομάτων των εκπροσώπων της επιχείρησης θα επιτρεπόταν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ακολουθήσει ενεργό προσέγγιση ε, τα ακούσατε σήμερα ε, τον διαμεσολαβητή που αναφέρθηκε. Ε, πόσο σημαντική αυτή είναι η προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό. Κάτι που απαιτείται και από του κανόνε για την προστασία των δεδομένων. Εκ των προτέρων αποσαφηνίζεται στου ενδιαφερομένου ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν δημόσια και ποια όχι. Εδώ και μερικέ εβδομάδε, τον Μάρτιο, δημοσίευσαμε ένα έγγραφο στην ιστοσελίδα μα εξηγώντα τι σημαίνει αυτή η ενεργό προσέγγιση λεπτομερέστερα. Το έγγραφο δείχνει ότι σε περιπτώσεις όπου η δημόσια αποκάλυψη των δεδομένων δικαιολογείται, αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει το ότι αυτή η αποκάλυψη είναι νόμιμη και δίκαια και ότι τα στοιχεία ο ενδιαφερόμενο ενημερώνεται πλήρω και μπορεί να απολαύσει των δικαιωμάτων του γιατί που απορρέωνε του δεδομένων. Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πολιτών, έτσι, τα συμφέροντα εκείνου που ζητά τι πληροφορίε, εκείνου το οποίο οι πληροφορίε αποκαλύπτονται και τέλο και τα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έτσι είναι αποτελεσματικότερη διαδικασία. Και ακούσαμε επανειλημμένε αναφορέ σε προβλήματα ε, προσωπικού. Μία ενεργό τέτοια ε, προσέγγιση μειώνει το γραφειοκρατικό άχθος και μειώνει τις επιπλοκές που ακολουθούν αιτήματα όπως την υπόθεση Bavarian Lager. Στο έγγραφο ενθαρρύνουμε τη δίκηση να αναπτύξει πολιτικές όσον αφορά αυτή την ενεργό ε, προσέγγιση. Ε, είναι σωστή εξισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων. Διαμορφώνται τις πολιτικές, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται επικοδομητικά το ένα με το άλλο και να ανταλλάσσουν τις πρακτικές σχετικό με τη σημερινή συζήτηση είναι και κάτι άλλο. Ότι το παρόν νομικό πλαίσιο δεν προσφέρει επαρκείς ουσιαστικούς προσανατολισμούς για τις περιστάσει κατά τι οποίες η ισορροπία των διαφόρων συμφερόντων γενικά είναι υπέρ τη αποκάλυψης. Δηλαδή, τα θεσμικά όργανα δεν γνωρίζουν ποιο επίπεδο διαφάνεια δικαιολογείται σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Και καμιά φορά οδηγούν σε, οδηγούνται σε αντανακλαστικό που δεν βοηθά ω αντίδραση. Το λέμε αυτό υπέρ τη ασφάλεια δικαίου. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει. Και ακριβώ, αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ προσετέθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού όταν υιοθέτησε την τροπολογία στην Ολομέλεια του Μαρτίου 2009 σχετικά με αυτό. Αυτή η τροπολογία επανεμφανίστηκε σε σχέδιο εκθέσεω τη Επιτροπή σα πέρσι το Μάιο. Αυτή η τροπολογία παρέχει τους αναγκαίους προσανατολισμούς και διευκρινίζει ότι πρέπει καταρχήν, μάλλον καταρχήν η σωστή ισορροπία είναι υπέρ της αποκαλύψεως στοιχείων αν τα στοιχεία αφορούν μόνο την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου εν γέννη δηλαδή. Αν τα στοιχεία αποκλειστικά σχετίζονται με δημόσιο πρόσωπο που δρά βάσει των, αυτής της ιδιότητας ή αν έχουν δημοσιευθεί ήδη τα δεδομένα με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Ε, υποστηρίζουμε πλήρω τι τροπολογίε που θετήθηκαν από το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ειλικρινά αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εν γέννη να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο στι συζητήσει που ε, θα ακολουθήσουν. Με ενδεχόμενη υιοθέτηση τη πρόσφατη προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή θα γραμμιστεί ο κανονισμό 1049 με τι απαιτήσει τη συνθήκη Λισαβόνα, η νομική αναγκαιότητα τη γενική αναθεωρήσεω ίσω να μειωθεί. Όμω παρόλα αυτά θα έλεγα υπάρχει ηθική και πολιτική αναγκαιότης να διευρυνθεί το παρόν πλαίσιο και για τη συμφιλίωση των κανόνων για την πρόσφαση του κοινού στα έγγραφα με τις ανάγκες προστασία των δεδομένων. Σας προσφέρω βοήθεια αν χρειαστείτε για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες για επαλήθευση φερρυπίν κατά πόσο οι προτινόμες τροπολογίες εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις. Μην διστάσετε αν θέλετε πληροφορίες να έρθετε σε επαφή μαζί μας, εάν χρειαστείτε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Uh, ε, θα κλέψω μερικά λεπτά από το τέλος της ε, συνάντησης για να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, στους ε, δύο προηγούμενους ομιλητές, ε, την καθηγήτρια κ. Κάρτιν και τον κ. Χέστινγκς. Ε, ήθελα να πω ότι ήταν τόσο εξαιρετική η παραφετηρή του που ήδη έδωσαν απαντήσει στι ερωτήσει που είχαν δημιουργηθεί, αλλά βλέπω ότι η κυρία Χαουτάλα κάτι έχει να πει. Κύριε Χάστινγκ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα και οι προτάσει σα για το πώ η νομοθετική διαδικασία του κανονισμού θα έπρεπε να συνεχιστεί. Ε, μια, Ίσως θα έπρεπε να πούν δύο λόγια και ο κύριος Διαμαντρούς και η κυρία Κέρτιν, γιατί εμείς ως, ε, ε, ε, κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς επιλογές μας για το πώς θα χειριστούμε τις προτάσεις της Κομισιόν που διευρύνουν το πεδίο του κανονισμού. Πώς να χειριστούμε αυτές τις δύο προτάσεις. Ε, η κυρία Χαουτάλα νομίζω απευθύνει την ερώτηση σε τρία άτομα, αλλά δίνω το λόγο καταρχήν στην κυρία Κέρτιν. Στις δύο προτάσεις πώς θα απαντήσετε την αναδιατύπωση του 2008 και την καινούργια πρόταση της Κομισιόν. Πώς να χειριστούμε αυτές τις δύο προτάσεις. Κυρία Κόρτιν, νομίζω ότι είναι πολύ ε, δύσκολο. Η πιο πρόσφατη ε, είναι διακοσμητικής φύσεως. Αναφέρει μόνο αυτά που λέει η συνθήκη έτσι κι αλλιώς ε, με έναν τρόπο έτσι πιο ρητό στον κανονισμό. Οπότε προσωπικά να σας πω το εξής υπό το φως των διευκρινήσεων που έχουν δοθεί και από την νομολογία και από την ίδια την συνθήκη και, την, και τη χάρτα ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αναδιατύπωση του κανονισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ε, η, τελευταία πρόταση θα μπορούσε να λείπει κιόλας τελείως. Ο ε, κύριος Χάστινγκς. Ε, ναι, και τα δύο. Όχι το ένα είτε το άλλο και τα δύο. Ε, το πεδίο εφαρμογή, ε, εντάξει, καλοδεχούμενο, ε, επικαιροποιεί το κείμενο, αλλά το θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο να ενταχθεί στην πρόταση αναδιατύπωσης. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να συνεχίσει το δρόμο της και αυτή η πρόταση. Κ. Διαμαντούρος, συμφωνώ απόλυτα η ιδέα της τελευταίας πρότασης της ε, Κομισιόν είχε προταθεί και από μένα τον ίδιο στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Κάποια πολύ απλά πράγματα για να ε, προσαρμοστούμε στη συνθήκη στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα έτσι ώστε όλα τα όργανα υπηρεσίες και ε, οργανισμοί θα περιλαμβάνονται και θα καλύπτονται από το 1049. Για να μην καθυστερήσουμε δηλαδή το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση και στα έγγραφα αυτών των σωμάτων. Απ' την άλλη μεριά όμως χρειάζεται να προωθεί και η αναδιατύπωση. Ο κ. Κάσμαν, το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τη θέση του στα ψηφίσματά του και η προσέγγιση δική μου και της Επιτροπής από την άλλη μεριά είναι να γίνει μια βαθιά σε βάθος αναθεώρηση του 1049 λαμβάνοντας υπόψη και την ομοθεσία, την ομολογία συγγνώμη. Ε, κάτι που με οδηγεί στον επόμενο μιλητή μας. Όπως έχουμε, έχουμε πει συχνά ότι ο 1049 επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς θα δώσω το λόγο στον Βαλέριο Πλάκο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικός σύμβουλος εκεί και θα μας μιλήσει για την διαφάνεια σε μη νομοθετικές δραστηριότητες ή για οτιδήποτε άλλο θέλει να μας μιλήσει. Α, υπό την ότι θα ξεπεράσει τα 10 λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν μου επέτρεψα να επιλέξω εγώ τον τίτλο ε, της ε, προσέγγισής μου Τη παρέμβασή μου, αλλά μου είπα να μιλήσω όποια γλώσσα θέλω. Οπότε θα μιλήσω γαλλικά. Στο συγγνώμη με αυτού πρέπει να χρησιμοποιήσουν ακουστικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή που προκάλεσε τον κύριο προσκάλεσε τον κύριο Γκριφιέ που μου ανέθεσε να τον εκπροσωπήσω. να σας παρουσιάσω ποιο είναι το ιδιαίτερο καθεστώς της πρόσβασης στα έγγραφα, το καθεστώς που εφαρμόζεται στην ε, ε, δικαστική δραστηριότητα του οργάνου μας. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς λοιπόν το οποίο αναγνωρίζεται από το άρθρο 11 παράγραφος 3 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμα και πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνα το δικαστήριο δεν υπόκειτο στους κανόνες διαφάνειας και πρόσβασης στα ε, έγγραφα του 200, το άρθρο 255 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ε, σήμερα όμως υπόκειται σε τέτοιους κανόνες το δικαστήριο μόνο όμως όταν ασκεί διοικητικές δραστηριότητες. Η συνθήκη Λισαβόνα επιβεβαιώνει λοιπόν ότι το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των διοικητικών του δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, ε, υπόκειται στους ε, κανόνες πρόσβασης, ε, κοινής πρόσβασης στα έγγραφα ε, κάτι το οποίο ε, αντικατοπτρίζεται και στις ε, πρόσφατες προτάσεις Κομισιόν για τροποποίηση του 1049 που αντιγράφουν ακριβώς την διατύπωση της συνθήκης Λισαβόνας που εξαιρεί το, Ευρωπαϊκό, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από, την, από τους κανόνες του 1049 όταν ασκείται αρμοδιότητες μη διοικητικής φύσεως. Συνεπώς, ε, σε αυτές τις δραστηριότητες διεπόμαστε από ε, τις, τους δικούς μας εσωτερικούς κανόνες και από ε, τις δικαιοδοσίες οι οποίες μας έχουν χορηγηθεί. Οπότε είναι, ποιες είναι οι αρχές, το δικαίωμα πρόσβασης ισχύει μόνο για τα, τους διαδίκους ε, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα σε πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις, τα δικόγραφα. Υπό την προπόθεση δεν υπάρχει, ε, ε με δύο προϋποθέσεις μάλλον, θα πρέπει πρώτον να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ε, της, ε, των σύσκεψης των δικαστών και να γίνονται σεβαστά τα προσωπικά δικαιώματα τα προσωπικά ε, δεδομένα. Συγγνώμη. Ε, ε υπάρχουν ε, έγγραφα τα οποία είναι διαβαθμισμένα και ενδεχομένως οι διάδικοι δεν θα έχουν πρόσβαση. Ε, τώρα, πλευράς κοινού. Τι πρόσβαση έχει το κοινό και οι κανόνες που εφαρμόζονται από τον εσωτερικό κανονισμό προβλέπουν ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρον μπορεί ε, να ε, συμβουλευτεί το ε, μητρό, το πρωτόκολλο δηλαδή. Αλλά όχι τα ίδια τα έγγραφα. Το κοινό έχει πρόσβαση στην ομολογία του δικαστηρίου, δηλαδή τις αποφάσεις που δημοσιεύονται ε, επί τη βάση δυνάμει ε, ε, των υποχρεώσεων του, του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που φορτώνονται στον ιστότοπο του δικαστηρίου στον οποίο έχουν άμεση πρόσβαση οι πολίτες. Απ' την άλλη μεριά στο πλαίσιο του σεβασμού της ανωνυμίας και των ε, απόρριτων πληροφοριών υπάρχουν και εκεί περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού. Μετά από ε, άδεια του Πρόεδρου, ε, ή του Πρόεδρου του Τμήματος, ε, είναι δυνατόν να δοθεί πρόσβαση ε, σε ένα τμήμα της ε, δικογραφίας μιας υπόθεσης σε τρίτους υπό την προπόθεση ότι αυτοί οι τρίτοι θα δικαιολογήσουν ε, το, τα ένομα συμφέροντά τους. Ε, και είναι δυνατόν αυτός ο οποίος θα λάβει την απόφαση να ακροαστεί ε, τους ενδιαφερόμενους. Είναι μια δυνατότητα όμως αυτό, δεν είναι υποχρέωση. Είπαμε ότι το δικαστήριο δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις διαφάνειας, ε, στις μη διοικητικέ ε, υποθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα δικόγραφα τα σχετικά με τέτοιου είδους ε, διαδικασίες εξαιρούνται. Τι εννοώ, αναφέρομαι στην απόφαση του Σεπτεμβρίου 2010 Σουηδία εναντίον Κομισιόν ε, εκεί το δικαστήριο είπε το εξής. Το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις διαφάνειας δεν αποκλεί την περίπτωση ο ένας πολίτης να έχει πρόσβαση σε έγγραφα ε, τα οποία έχουν σχέση με μια υπόθεση υπό την προπόθεση ότι αυτή η αίτηση έχει υποβληθεί σε άλλα όργανα και όχι στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για αιτήματα τα οποία υποβάλλονται κατευθείαν, απευθείαν σε άλλο ε, όργανο και όχι στο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, κατέχει τα ειδικόγραφα. Ε, ένα, μια αίτηση πρόσβαση σε τέτοιου είδου ε, έγγραφα θα πρέπει να την χάνει χειρισμού στο πλαίσιο του κανονισμού του 1049 και να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις που προβλέπει ο 1049 στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Δύο λεπτά ακόμα έχετε, λέει ο πρόεδρο. Δύο στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την προστασία αυτή. Ε, ε, η, υποχρέωση καλής ε, ε απόδοση δικαιοσύνης και το δικαίωμα των διαδίκων να ε, διατηρούν το απόρριτο των ε, σκέψεών τους. Ε, πάση περιπτώσει αυτή η διαδικασία αφορά αυτές οι εξαιρέσεις, δηλαδή αυτός ο περιορισμός αφορά μόνο εκκρεμείς υποθέσεις, όχι τελε, υποθέσεις που έχουν τελεσυδικήσει ή έχουν εκδικαστεί. Ε, αυτό το τεκμήριο δεν υπάρχει πλέον όταν η υπόθεση έχει κλείσει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ε, να ε, εξετάζουμε, μάλλον θα πρέπει να εξετάζουμε κατά περίπτωση να αν υπάρχει θέμα βλάβης αυτών των συμφερόντων. Η, το, ε, το Συμβούλιο προσέφυγε πρόσφατα στο δικαστήριο για ένα θέμα ε, δικογράφων από κράτη-μέλη που υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένη υπόθεση ε, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον η υπόθεση έχει κλείσει ε, δεν υπήρχε θέμα προσβολής ή βλάβης των δικαιωμάτων του κράτους μέλους συνεπώς το δικαστήριο έδωσε την σύμφωνη γνώμη του για την δημοσιοποίηση των εγγράφων. Μπορώ να σταματήσω εδώ αλλά είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.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 Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα και ο χρόνο που αφιερώνουμε δεν είναι επαρκή. αλλά ζητώ συγγνώμη από όλου του ομιλητέ που του ζητώ να είναι σύντομοι. Τώρα έχουμε τον κύριο Αλφρέντο Παρανέλα, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι υπεύθυνο τη ε, μονάδα ε, που ασχολείται με την ε, σωστή διαχείριση δημοσίου χρήματο. Κάτι που μα ενδιαφέρει όλου. Κύριε Παναρέλα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω και εγώ τον κανόνα των δέκα λεπτών. Έχω την τιμή σήμερα να σας παρουσιάσω τη δική μας προσέγγιση για την πρόσβαση στα έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άρχισε να δίνει πρόσβαση στα έγγραφα από το 1997 όταν υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά αυτοί οι κανόνες από τα διοικητικά μας όργανα. Η πρόσβαση, η πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήταν περιορισμένη εκείνη την εποχή. Οι κανόνες ε, του 1997 αναθεωρήθηκαν το 2002 μετά τον κανονισμό 1049 για να ανταποκρινόμεθα στις ε, ε, διατάξεις και όλα τα όργανα θα έπρεπε να έχουν εσωτερικούς κανόνες για την πρόσβαση και πρόσβαση στα έγγραφα και γνωστοποίηση το 2006, το 2007 και το Φεβρουάριο του 2010 τροποποιήθηκαν εκ νέου οι κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα που έχουμε και τώρα αποκαλούνται πολιτική διαφάνεια στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων ε, Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες ε, τις ε, ε, διατάξεις που ισχύουν και τη Σύμβαση Όρχους και την νομοθεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης του Όρχους στα κοινοτικά όργανα. Ο κανονισμός 1049 εφαρμόζει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά την άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων ε, και αυτά τα οποία έχουν σχέση με το άρθρο 15 της συνθήκης, αλλά η πολιτική διαφάνεια της τράπεζας προχωρεί πολύ περισσότερο και το κείμενο της πολιτικής διαφάνειας μας ε, ε, τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού 1049. Η πολιτική ε, διαφάνεια της Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, είναι ότι τηρούμε τους κανόνες περί εκτός εάν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Η τράπεζα θα πρέπει να διαφυλάσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όσον αφορά στοιχεία των πελατών της χρηματοδοτών και επενδυτών και εξετάζουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν επιπτώσει ε, στα συμβαλλόμενα μέρη και που ε, μπορεί να εμποδίζει την τράπεζα από την υλοποίηση των στόχων της. Θα αρνηθούμε λοιπόν την πρόσβαση στα δεδομένα όταν ε, τίθεται σε κίνδυνο εμπορικά συμφέροντα, πνευματική ιδιοκτησία η εσωτερική απόλυτη διαδικασία της ε, τράπεζας. Είναι οι, ίδιε ίδιες δηλαδή, που υπάρχουν και στον κανονισμό 1049. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, μπορεί να δίνει στοιχεία σχετικά με ε, τα συμβαλόμενα μέρη μας, με τους χρηματοδότες και πελάτες και μπορούν όλοι να ζητούν πληροφορίες από την τράπεζα και όταν η τράπεζα εξετάζει αίτημα για πληροφόρηση δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη προτεραιότητα η τράπεζα σε συγκεκριμένα αιτήματα χορήγησης πληροφοριών. Υπάρχει και ένας επίσημος μηχανισμός ε, παραπώνων, ένας επίσημος ε, ε, μηχανισμός που υπόκειται στο Γενικό Γραμματέα για, την, ε, για τις καταγγελίες και διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι μια εσωτερική διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε προσφυγή στον διαμεσολαβητή. Δεν προδικάζει την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η διαδικασία αρχικά περιορίστηκε σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή όμως η ΕΤΕΠ έχει λειτουργήσει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να καλύψουμε τις δυνατότητες για πολίτες που δεν είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μας, έχουμε μία συμφωνία, ένα προσύμφωνο με τον διαμεσολαβητή και του αναθέτουμε ε, ε, το έργο να λαμβάνει καταγγελίες και από πολίτες που δεν είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτονται όλοι οι συμβαλόμενοι με εμά. Η ΕΤΕΠ ως νέος οργανισμός έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόζει το ύψιστο επίπεδο διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητε της και το θεωρούμε τμήμα τη αποστολή μας και τμήμα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να εκπληρώνουμε. Η ΕΤΕΠ κάθε τρία χρόνια οφείλει να αναθεωρεί τις αρχές της περί διαφάνειας, ούτως ώστε να επικαιροποιούμε ε, αυτά τα οποία ισχύουν βάσει των όσων ισχύουν στον κλάδο. Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και σε σχέση με άλλους ε, φορείς η πολιτική της ΕΤΕΠ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλές επιτροπές ε, παρακολουθούν την πολιτική διαφάνεια της ΕΤΕΠ και πολλές φορές μας έχουν κάνει χρήσιμες συστάσεις. Με βάση την έκθεση του κυρίου Κούτο, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο πέρασε ένα ψήφισμα το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα αυτή τη παρακολούθηση τη πολιτική τη ΕΤΕΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικέ προ όφελο των πολιτών και ακριβώ αυτό προσπαθούμε και εμεί να διασφαλίζουμε στην ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναρέλα. Τηρήσατε και το χρονοδιάγραμμά σας, αλλά και τελειώσατε και πιο νωρίς. Μας εξοικονομήσατε κάποια λεπτά πρέπει να χειριστώ με ευελιξία το θέμα. Πρέπει να έρθουν άλλοι τρει. Αλλά θα πρέπει και τα μέλη του πάνελ να είναι εδώ για να απαντήσουν και σε ερωτήσει. Ε, λάμπει πάντα η εξυπνάδα. Λοιπόν, θα ακούσουμε για δίποτε, δίποτε ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες τώρα, ερωτήσεις σχόλια και μετά θα τους αφήσουμε να φύγουν και θα έρθουν τα άλλα μέλη του πάνελ. Έχετε ερωτήσεις, έχετε σχόλια. Ορίστε. Ερώτηση για τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για τα δικαστηρία. Πώς ερμηνεύεται το διοικητικό καθήκον σύμφωνα από τη συνθήκη τη Λισαβόνα για τη δικαστήρια και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν κατάλαβα καλά πώς θα εφαρμόσετε τη σχετική διάταξη. Λέτε ότι οι κανόνες σας περί προχωρούν πιο πέρα από το άρθρο 15 της συνθήκης. Πρόεδρος, μπορείτε να μας πείτε ποια διάταξη. Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Α, πώς ερμηνεύεται το διοικητικό καθήκον που αναφέρεται στο άρθρο 15 της συνθήκης που λέει ότι ο κανονισμός θα ισχύει στο δικαστήριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο όταν ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο για μας, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και θα με ενδιαφέρε να γνωρίζω πώς ερμηνεύουν τη σχετική διάταξη για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είπατε ότι οι κανόνες περί προχωρούν πιο πέρα από το άρθρο 15 της συνθήκης και ότι τηρείται τον κανονισμό. Αλλά σε οδήποτε έτοιμα υποβάλλουμε, μας υπενθυμίζετε ότι ο κανονισμός ισχύει μόνο σε εσά όταν ασκείτε διοικητικό σας καθήκον. Πολύ καλό νομικό ερώτημα, με πολλές πολλές απαντήσεις, φοβάμαι. Μπορούμε να σας στείλουμε αναφορά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Τάπεζα Επενδύσεων και όπως προαναφέρατε στην παρουσίασή σας, αν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις του κανονισμού δεν μπορείτε να τους κατηγορείτε αυτούς αλλά τον κανονισμό. Γι' αυτό γίνεται αναθεώρησή του. Δεν σας ξαναδώσω το λόγο, διότι είστε νομικός και θα το χρησιμοποιήσετε πολύ καλά το χρόνο. Λοιπόν, πρώτα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά ο συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα απαντήσει. Για τα διοικητικά καθήκοντα, απλούστατα, ε, έχει δρομολογηθεί η προσπάθεια, το εγχείρημα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει εργασίε. Ερχόμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε το άρθρο 15 περί διοικητικών καθηκόντων. Ακόμα εξετάζουμε το θέμα. Εκρεμεί. Για τα άλλα σημεία. Με εκπλήσει αυτό που λέτε ότι απορρίπτουμε τα αιτήματά σας. Δεν είπα κάτι τέτοιο λέει κυρία. Δεν θα αρχίσει συζήτηση, λέει ο κύριο Κάσμαν, για ένα αίτημα, ε, για κάποια αιτήματα συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργανώσεω. Ευχαριστώ ο συνάδελφο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το μελετούμε το θέμα στα πλαίσια της εγκρίσεως του εσωτερικού κανονισμού. Δεν μπορώ να προβλέψω τις εκτιμήσεις που θα γίνουν επί του θέματος. Προσωπικά μπορώ να πω ότι οι διοικητικές λειτουργίες αφορούν θέματα προσωπικού, εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού των κοινοτήτων, τίθεται διάφορα θέματα, όπως δημόσιες προμήθειες, οι οποίες καλύπτονται από αυτή την έννοια που αναφέρεται εκεί με κάποια ενδεχόμενη εξαίρεση ε, για την προστασία κάποιων συμφερόντων ενδεχομένω. Όπως είπατε λέει ο Πρόεδρος με την επιφύλαξη βεβαίως των περαιτέρω αποφάσεων και ανακοινώσεων. Κύριε Διαμαντούρο, έχετε κάποιο σχόλιο. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κάτι που σχετίζεται με αυτό που είπε ο κύριος Χέστινγκ για την ενεργή προσέγγιση. Είναι στο επίκεντρο αυτή η δραστηριοποίηση της ουσίας του κανονισμού. Α, όπως ερμηνεύω τουλάχιστον τη θέση και του Κοινοβουλίου. Θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν αυτό το θέμα. Ζητείτε από τα θεσμικά όργανα να σκέφτονται εκ των προτέρων, να προβλέπουν όταν ετοιμάζουν τα εγγραφά και να εντάσσουν στα έγγραφα τη δυνατότητα σύμφωνα με την οποία θα ζητηθεί πρόσβαση και να αποφευθεί να γίνεται κάτι τέτοιο εκ των υστέρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι που θέλω να φέρω δημοσία. Η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το γνωρίζει. Και Ήθελα να του συγχαρώ, ε, διότι ε, το μήνυμα δεν το έχουν εστερνιστεί κάποιε γενικές διευθύνσεις. Τόσο αφορά το δικαστήριο, να πω απλώς ότι το δικαστήριο έδωσε πάρα πολύ σημαντικούς προσανατολισμού όσον αφορά τη συγκεκριμένη επακριβή ερμηνεία πολλών από αυτές τις διατάξεις και πρέπει να γίνει αυτό κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, όσον αφορά τις θέσεις των κρατών μελών. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Σουηδία και για άλλε περιπτώσει. Αν το ξεκαθαρίσετε αυτό, θα μα βοηθήσετε πολύ για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εγώ, σαν διαμεσολαβητή, θέλω να καταγραφεί ότι λέγω ότι επί της Προεδρία του κ. Μέιστατ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άλλαξε πορεία. Ήταν ένα θεσμικό όργανο που έλεγε συγγνώμη, είμαστε μια τράπεζα. Ε, δεν μπορείτε να μας υποχρεώσετε να είμαστε πολύ προσβάσιμοι. Και τι έγινε τώρα, άλλαξε. Και λέει τώρα είμαστε τράπεζα, αλλά είμαστε και ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, άρα είμαστε υπόλογοι, άρα πρέπει να λογοδοτούμε, άρα πρέπει να δίνουμε πρόσβαση στι πληροφορίε μα. Και ήταν άκρο θετικέ οι επαφέ μα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάσει αυτού. Επί τη βασική υποθέσεω ότι τελικά οι πληροφορίε θα είναι διαθέσιμε. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσει. θα ζητήσω από τα νέα μέλη του πάνελ να έρθουν. Είναι εκπρόσωποι της Frontex, της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Και παρακαλώ να ευχαριστήσετε τους συμμετέχοντες που αποχωρούν τώρα από το έδρανο. Και τώρα το τελευταίο τμήμα για τη διαφάνεια στις υπηρεσίες στους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε εκπροσώπους της Frontex, της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής της νομικής μονάδας της Frontex. Σακχάρη Βουραλουνσόλο είμαστε φρικτοί οι Βρετανοί στην προφορά και έτσι αυτή είναι η εικόνα που δίνουμε και τελικά εγώ συμμορφώθηκα με τα στερεότυπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχεδόν δύο θέα. Βούρεν σολάιστε, έπρεπε να το πείτε. Δεν με πειράζει όμως, δεν πειράζει. Ξέρω ότι πρέπει να βιαστώ, δεν έχω πολύ χρόνο. Σας πω μερικά λόγια για τη Frontex, διότι υποθέτω ότι πολλοί από εσά δεν γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Η Frontex είναι ένας οργανισμός Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει σαν καθήκον να συντονίζει και να διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς ελέγχου των συνόρων των κρατών μελών να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένα από τα αποτελέσματα του κεκτημένου Σέγγεν, όπως αποκαλείται, της συνεργασίας Σέγγεν. Δηλαδή, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να έχουν παρόμοιο επίπεδο, υψηλό επίπεδο ελέγχου. In order to facilitate that. Και δημιουργήθηκε η Frontex για να το διευκολύνει αυτό, να συντονίζει τι κοινέ δραστηριότητε των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτά που είχα να πω στην αρχή τώρα περί διαφανείας ή προσβάσω στα έγγραφα. Ο κανονισμός της Frontex, ο κανονισμός που δημιούργησε τη Frontex, ε, είναι πολύ σύγχρονος κατά την άποψή μου. Υιοθετήθηκε το 2004 και λέει ότι η υπηρεσία της Frontex μπορεί να κοινοποιεί στο κοινό κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας με γρήγορο, αξιόπιστο, εύληπτο τρόπο τις δραστηριότητές μας. Ε, υπέχουμε υποχρέωση σύμφωνα τον κανονισμό, σύμφωνα τον οποίο μπορούμε να κοινοποιούμε. Άρα στην πράξη υιοθέτησε η Frontex, αν μπορώ να το πω, αυτή την ενεργό, τη δραστήρια πολιτική ε, επικοινωνίας, μια από τις μονάδες μας, Ήδη του 2005 η πρώτη που δημιουργήθηκε αφορούσε την ενημέρωση του κοινού. Οπότε έχουν προσλάβει συγκεκριμένα άτομα ακριβώς γι' αυτό, για να προβαίνουν σε ανακοινώσεις τύπου, να ανακοινώνουν με εύληπτο τρόπο το τι κάνουμε. Το άρθρο 26 λοιπόν του κανονισμού μας λέει ότι η Frontex υπόκειται στον κανονισμό 1049. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε τον 10, ότι ο 1049 είναι ένας κανονισμός που αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, δεν αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες. Συνεπώς, η υποχρέωσή μας να κοινοποιούμε ε, ενεργά είναι ευρύτερη. Όμως, το θέμα μας εδώ είναι ότι ο 1049 πλαισιώνει την πρόσβαση στα έγγραφα. Οι πρόσβαση πληροφορίες ε, δεν ρυθμίζεται τόσο από αυτό το άρθρο, αλλά από τον κανονισμό της Frontex. Λέει ότι δύναται να κοινοποιεί, ενδέχεται να κοινοποιήσει η Frontex. υιοθετήσαμε ή το Διοικητικό Συμβούλιο το 2006 υιοθέτησε απόφαση εσωτερική που καθορίζει λεπτομερέστερες διευθετήσεις περί της εφαρμογής του 1049. Αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύντομα θα ενημερωθεί, θα επικαιροποιηθεί λόγω των νέων αναγκών και των εξελίξεων και κυρίως λόγω του ενδεχομένου ενός νέου κανονισμού, αυτού που συζητούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα μας δώσετε και θα μας δείξετε καλά αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, θα ενημερώσουμε και εμείς τους, τον εσωτερικό μας κανονισμό. Κάποια λόγια για τις αιτήσει του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα της Frontex. Ελάχιστες τις αιτήσει έχουμε λάβει. Δεν το λέω γιατί θα ήθελα να μας ζητήσετε τα έγγραφά μας, αλλά έχουμε και ελάχιστους πόρους. Ίσως όμως αυτό οφείλεται στην ενεργή μας πολιτική, στη δραστηριοποίησή μας όσον αφορά την επικοινωνία. Έχουμε περίπου 10 αιτήσει το χρόνο για πρόσβαση στα εγγραφά μας, άρα δεν έχουμε πολλές αιτήσει όμως. Έχουμε μία πλήρη διαδικασία για αυτούς τους σκοπούς. Τώρα μερικές πρακτικές εμπειρίες μας. Όσον αυτό το θέμα, παρόλο που δεχόμαστε 10 αιτήσει το χρόνο, εν γέννη, οι υποχρεώσει που απορρέουν από τον κανονισμό 1049 δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα για την Frontex. Όμως υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα σημεία τα οποία ίσως θα συζητήσουμε. Το πρώτο για την πρόσβαση, ο κανονισμός αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και όχι στις πληροφορίες. Όμως, οι περισσότερες από τις δέκα ετήσιες εκθέσεις που λαμβάνουμε, ε, αιτήματα μάλλον που ε, δεχόμεθα, είναι αιτήματα για παροχή πληροφοριών. Πληροφορίες για αριθμό παρανόμων μεταναστών ή ε, αριθμό ετούντων άσυλο, ή ε, για κάποια διακίνηση που διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα. Ε, δεν αναφέρονται αυτά σε κάποιο έγγραφο. Πρέπει να κάνουμε εσωτερικές έρευνες και μελέτες για να απαντήσουμε και να θέσουμε τις απαντήσεις επί χάρτου και να στείλουμε κάποιο έγγραφο. Είναι κάτι παραπάνω από πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι αίτηση για πρόσβαση σε πληροφορίες. Δεύτερο σημείο που συζητήθηκε είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα κράτη-μέλη η Frontex διευκολύνει και συντονίζει τα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό ότι οι δραστηριότητές μας βασίζονται κατά πολύ επί της εμπιστοσύνης των κρατών μελών έναντι της Frontex. Ε, λαμβάνουμε πολλά έγγραφα και πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και πραγματοποιούμε πολλές αναλύσεις κινδύνου όσον αφορά απειλές και κινδύνου στα εξωτερικά σύνορα για αυτές τις αναλύσεις περί απειλών το υλικό προέρχεται κυρίως από τα κράτη-μέλη. Και αυτό το υλικό είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα κυρίως. Τα κράτη-μέλη λοιπόν... Α, είχαμε κάποιες ερωτήσεις από κράτη-μέλη, κάποιες αιτήσεις από κράτη-μέλη για πληροφορίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό πάμε στα κράτη-μέλη και ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους και συνήθως τα κράτη-μέλη δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά το σύστημά μας. Δεν ομά, όχι όταν μη δίνετε τι πληροφορίε. Όταν μα ζητάνε να δώσουμε πληροφορίε που μα δώσανε τα κράτη-μέλη, λένε όχι. Μην τι δίνετε. Και εγώ προσπαθώ σαν νομικό σύμβουλο να πείσω τα κράτη-μέλη. Ναι, έχετε δυνατότητα αρνησή κυρία, αλλά θα πρέπει να ε, δώσετε ένα λόγο, κάποιο ε, αίτιο. Ε, μια αιτιολογημένη απάντηση γιατί δεν πρέπει να δώσουμε ένα έγγραφο που μα στείλατε. Αυτό είναι κάτι που ελπίζω μπορεί να το ρυθμίσει ο νέο κανονισμό και να μα βοηθήσει. Τρίτον, σημείο, είναι μερική απελευθέρωση εγγράφων, δηλαδή να διαγράφουμε κάποια τμήματα ενός εγγράφου το οποίο στέλνουμε. Πολύ συχνά μας ζητούν να τους πούμε ποια είναι τα επιχειρησιακά μας σχέδια ή ποιες είναι οι εκθέσεις αξιολογήσεώς μας. Είναι μακροσκελή έγγραφα. Έχουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες σελίδες. Και τα περισσότερα έγγραφα κάπου συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που λάβαμε από κράτη-μέλη και που θεωρούνται πιστευτικές. Μερική διάθεση εγγράφων σημαίνει πολύ διοικητική δουλειά για μας. Πρέπει να εξετάσουμε το έγγραφο σελίδα προς σελίδα, να κάνουμε διαγραφές εδώ και εκεί. Οπότε εδώ είναι το θέμα της αναλογικότητας και του διοικητικού άχθους που τίθεται. Όμως ε, βρήκαμε μια νέα λύση που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε με ενεργό τρόπο πάντα. Ήδη εκ των προτέρων εμείς ετοιμάζουμε εκθέσεις αξιολόγησης. Εκθέσεις αξιολόγησης των συντονισμένων επιχειρήσεών μας στα εξωτερικά σύνορα. Ήδη από την αρχή ετοιμάζουμε τη δημόσια εκδοχή του εγγράφου και την εσωτερική εκδοχή του εγγράφου. Και ελπίζω αυτό να βοηθήσει. Δηλαδή, όταν κάποιος ενδιαφέρεται για κάποια επιχείρηση, μπορούμε να του δώσουμε τη δημόσια εκδοχή του εγγράφου και εμείς κρατάμε μόνο κάποιες πληροφορίες για το εσωτερικό έγγραφο πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιους σκοπούς ή δημοκρατικούς σκοπούς, αλλά είναι στατιστικά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα των κρατών μελών ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες. Και βέβαια το τελευταίο που έχουμε εμπειρία, τα ευαίσθητα έγγραφα. Ξέρετε, άρθρο 9 του κανονισμού λέει αν φέτε στα ευαίσθητα έγγραφα. Τι είναι ευαίσθητο έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο έχει διαβαθμιστεί σύμφωνα με τους κανόνες εκείνου που ε, συνέταξε το έγγραφο. Όταν ο συντάκτης του εγγράφου το έχει διαβαθμίσει. Δεν έχουμε περιθώρια μεγάλα για λιγμούς. Το πρόβλημα ποιο είναι, και το είδα στην πράξη όταν έκανα τη δουλειά μου, ότι είναι τόσο εύκολη αυτή. Είναι πολύ εύκολη η διαβάθμιση του εγγράφου να γίνεται χωρίς να εξηγείται γιατί είναι μυστικό, είναι απόρριτο ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Ίσως ε, μπορεί εκεί να βρεθεί κάποια λύση στο μέλλον, να μας βοηθήσει. Δύο λεπτά μου έμειναν. Λοιπόν, εν γέννη, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την αναδιατύπωση του κανονισμού δεν δημιουργεί κάποια συγκεκριμένα προβλήματα για μας. Εξετάσαμε την πρόταση, δεν έχουμε πρόβλημα, συμφωνούμε και εδώ έχω παραθέσει κάποιους από τους ιδιαίτερους τομείς που μας ενδιαφέρουν ε, σχετίζονται με αυτά που προανέφερα Υπάρχει μια νέα εξαίρεση που σχετίζεται με την ασφάλεια φυσικών νομικών προσώπων. Θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τι σημαίνει αυτό για μας. Υπάρχει νέος λόγος για εξαίρεση αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία επιλογών διότι για συστήματα πληροφορικής και για μελέτες ε, προκυρήσουμε διαγωνισμούς, ε, πρέπει να το μελετήσουμε προσεκτικά. Τα μη εντοπίσιμα έγγραφα, το ίδιο αφορά για την πρόσβαση στα έγγραφα και την πρόσβαση στις πληροφορίες, αυτά που είπα, χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσει στο νέο κανονισμό, πληρωμές για τα έγγραφα που διατίθενται, ενδιαφέρουσα καινοτομία, ποτέ δεν ζητήσαμε χρήματα, δεν ξέρω. Τώρα την εποχή αυτή, τη δύσκολη οικονομικά, μπορούμε να το σκεφτούμε και σχέση με προσβάσεις του κοινού στα έγγραφα και προστασία ιδιωτικών δεδομένων, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Χέιστινγκς, είναι κάπως αφήσει η κατάσταση λόγω της πρόσφατης δικαστικής απόφασης. Ελπίζω και αυτό να διαλευκανθεί και να ξεκαθαριστεί στο εγγύ μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόρεν Σόλα για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ δεν θα μελετήσω λεπτομερώς αυτά τα οποία ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναδιατύπωσή του. Θα έλεγα περισσότερο να δώσουμε σημασία σε αυτά που προτείνει το Κοινοβούλιο, που είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που θα ήθελαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και όταν λέω Επιτροπή και Συμβούλιο εννοώ τα θεσμικά όργανα και όχι τα συγκεκριμένα άτομα που εργάζονται μέσα σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα σε μια παρέμβαση από τον επικεφαλής νομικών θεμάτων της Europol. Ο κύριος Ντίτριχ Νιούμαν έχει το λόγο. Thank you, Chair. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε. Είναι τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μια παρέμβαση PowerPoint που δεν θα διαρκέσει πάνω από λίγα λεπτά. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας καθώς και την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όταν θα εξετάσει τον κανονισμό να σας μιλήσω καταρχήν ε, για ε, μια επιχείρηση διάσωσης από το Μάρτιο του 2001 ε, που η αστυνομία συνέλαβε υπόπτους για κακοποίηση παιδιών. Εντοπίστηκαν πολλοί υποπτοί και τοποθετήθηκαν σε ασφαλή χώρο 232 παιδιά είχαμε πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία είχαν οι δράστες και εμπλέκονταν πάρα πολλά έγγραφα στην όλη αυτή τη διαδικασία, έγγραφα τα οποία υπόκειται βέβαια στις διατάξεις της οδηγίας. Πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη εμπιστεύονται την Europol και το λέω ως πρώην αστυνομικός αυτό, διότι συνήθως οι αστυνομικοί δεν εμπιστεύονται δεν έχουν εμπιστοσύνη σε ό,τι θα γίνει με τις πληροφορίες τις οποίες ε, διαχειρίζονται. τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε τις ε, φυλάσσουμε ε, σε χώρο στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες κατά την εργασία τους. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ η ορθή διαφύλαξη των πληροφοριών. Είναι καθήκον της Europol να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και μας ενδιαφέρει και το ποια είναι η αντιμετώπιση των αστυνομικών αρχών σε εθνικό επίπεδο έναντι των εγγράφων γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι εθνικές αρχές για τις οποίες επίσης οι λύσεις είναι πολύπλοκες. Το θέμα της λογοδοσίας και της ε, αρμοδιότητας της Europol όσον αφορά την ε, διαφάνεια νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε ως συνδεδεμένα θέματα. Εμείς ε, λογοδοτούμε προς τα θεσμικά όργανα της κοινότητας και προσφάτως τη Δευτέρα μόλις ήρθε ο κύριος Wainwright, διευθυντής της Europol ακριβώς για να περιγράψει τις δραστηριότητες μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. έχουμε ένα ε, υπεύθυνο προστασία των δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να λογοδοτούμε και προς το Κοινοβούλιο και προς την Επιτροπή και προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον είμαστε οργανισμό που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες τις οποίες δίδουμε προς τα κράτη-μέλη είναι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να γνωστοποιούνται και να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Είχαμε ένα καθεστώς ε, για την πρόσβαση στα έγγραφα και πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας και όταν ε, εγκρίθηκε η νέα νομική μας βάση είχαμε προχωρήσει σε μια αναδιατύπωση των κανονισμών που είχαμε για την πρόσβαση στα έγγραφα. Ε, τώρα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και σε μεγάλο βαθμό ακολουθούμε τον κανονισμό 1049. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1049, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της Europol και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα συστήματα ε, δεδομένων μας, παρότι αυτά αποτελούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. για άρνηση γνωστοποίηση, οι λόγοι που χρησιμοποιούμε είναι οι ίδιοι που αναφέρονται και στον κανονισμό 1049. Είχαν υποβληθεί 29 ε, αιτήματα από το 2007 και μετά ε, και σε αυτά και σε αυτά δόθηκε η δυνατότητα γνωστοποίησης και μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις δεν ε, δώσαμε δικαίωμα πρόσβασης. υπάρχει ε, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και το δικαίωμα των πολιτών για ασφάλεια και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο. Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπόκειται στις διατάξεις αυτές μόνο όταν ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα. Θα έπρεπε να αναφέρεται ε, και η Europol που αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αναφέρεται. Το δικαίωμα ασφάλειας, ε, το οποίο ε, αναφέρεται και στο άρθρο 88 της συνθήκης που αφορά τη Europol είναι κάτι το οποίο πρέπει ε, να υλοποιείται υπό τη μορφή μιας δυνατότητας άρνησης πρόσβασης ε, στα έγγραφα όταν υπάρχει θέμα δημόσιας ασφάλειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα, ήταν, ε, θα μπορούσα να σας αναφέρω έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται για πιθανές επιχειρησιακές ενέργειες και έγγραφα που αφορούν άλλες δραστηριότητες της Europol εγώ μιλώ καθαρά ως κάποιος ο οποίος στην πράξη ε, εφαρμόζει αυτόν τον κανονισμό και ξέρω ότι είναι πολύ ευρύτερη η συζήτηση, αλλά εγώ μιλώ μόνο ε, για τα θέματα που μας αφορούν στην πρακτική εφαρμογή. Η εξαίρεση που χορηγείται είναι πάρα πολύ στενά εννοούμενη. εμείς πολλές φορές έχουμε συμφωνίες βάσει των οποίων δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων. το δικαίωμα των πολιτών για την πρόσβαση σε δεδομένα ε, πρέπει να εξισορροπείται με το δικαίωμα ασφάλειας των πολιτών. Εδώ επισέρχεται το παράδειγμα της υπόθεσης Bavarian Lager, όπου ε, δεν θα έπρεπε να υπονομεύεται η ασφάλεια ε, των εμπλεκομένων από την αποκάλυψη δεδομένων για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Έχουμε πάρα πολλά συστήματα δεδομένων, πάρα πολλά δεδομένα τα οποία ε, διαχειρίζεται η Europol και έτσι θα έπρεπε τα συστήματα δεδομένων της Europol να αποκλείονται, να εξαιρούνται από την ε, δημόσια πρόσβαση. Δηλαδή όλα τα έγγραφα της Europol, και μην βάλετε τις φωνές σε αυτά που σας λέω, ε, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του κανονισμού όταν θα συζητήσετε τον κανονισμό είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Επίσης δεν θέλουμε να δημιουργούνται νομικά και να έχει το δικό της σύστημα που επιτρέπει στον υποκείμενο στα δεδομένα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή τους. Η λογοδοσία λοιπόν και η προστασία των δεδομένων διασφαλίζονται μέσω αυτών. Ένα λεπτό μόνο έχετε στη διάθεσή σας ακόμη. Ξέρω είναι πολύ δύσκολο να ε, συντομεύσω. Είχα τρία σημεία και θα προσπαθήσω να αναφέρω μόνο τα δύο ή και ίσως το μόνο το ένα. Η γνωστοποίηση ονομάτων και ε, λειτουργιών στο πλαίσιο της δουλειάς της Europol είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα διότι υπάρχει δυνατότητα προστασίας ε, ε, ονομάτων, ιδίως για θέματα που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα να ε, αναφέρω κάτι ακόμη που είναι περισσότερο διοικητικού χαρακτήρα. Ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα τα οποία έχει ένας οργανισμός. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαιρούνται τουλάχιστον τα συστήματα δεδομένων της Europol διαφορετικά. Ε, συνεχώς θα βρισκόμασταν σε ε, αθέτηση του κανονισμού. Όπως και στο άρθρο 15 θα πρέπει να εξετάσουμε το αν οι υποχρεώσεις της Europol οφείλουν να περιορίζονται σε διοικητικά έγγραφα και μόνο έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μεμονωμένε επιχειρήσει ή με εξελίξει αστυνομικέ επιχειρήσει ή ακόμη και παρελθούσε αστυνομικέ επιχειρήσει, όπου και πάλι δεν μπορεί να υπάρξει γνωστοποίηση ε, και εδώ θα πρέπει να είναι περίπτωση εγγράφων τα οποία δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε ε, λίγο χρόνο παραπάνω. Ολοκλήρωσα εδώ την παρέμβασή μου. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είτε σε νυν σε πρώην αστυνομικό πάντοτε θα δίνω μερικά πρόσθετα δευτερόλεπτα. Ε, και οι συγητέ και η Επιτροπή προθύμω θα δεχτούν οποιαδήποτε γραπτή παρέμβαση θέλετε ε, να υποβάλλετε και εσείς και οποιοδήποτε ποτέ άλλος από τους παρεμβαίνοντες. Τέλος, Έχουμε την παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο λόγος στην ε, ε επικεφαλής του Γραφείου των Βρυξελών της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, την Ζωζιάν Ριβιέρ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε. Να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με μια σύντομη παρουσίαση της ε, υπηρεσίες μας και των δραστηριοτήτων της και μετά θα σας ε, ενημερώσω ε, την εμπειρία μας σε ό,τι αφορά τα θέματα πρόσβαση σε δικαίωμα ε, και σε θέματα πρόσβασης σε πληροφορίε για το περιβάλλον από πλευρά του κοινού όπως προβλέπεται τον κανονισμό του έρχους 1367-2006. Πρόκειται για δύο κανονισμού που καλύπτουν τους τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία ε, και στι πληροφορίε που προκύπτουν απορρέων από την ε, εντολή μα. Ε, είμαστε μια υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με έδρα την Κοπενχάγη, λειτουργούμε από το 1994. Αποστολή μας είναι να δίνουμε στου αυτούς που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις αλλά και στο κοινό τι πληροφορίε που είναι απαραίτητε, ανεξάρτητες, εστιασμένε και επαρκείς έτσι ώστε ε, να μπορούν να, να συνεισφέρουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Στην ε, διαδικασία επεξεργασία και υιοθέτηση τη κοινωνική νομοθεσία, η υπηρεσία μα ανταλλάσσει διάφορου διαφόρων ειδών έγγραφα, μελέτε, δεδομένα, δείκτε κλπ. με την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη τη ε, υπηρεσία μα που είναι 32 συγκεκριμένα, 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση και η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Τουρκία και η Ελβετία. Πέραν αυτού του βασικού πυρήνα των, πολιτικών ε, ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο, συνεργαζόμαστε με άλλα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Ευρωπαϊκή Οικονομική ε, και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ. Επίση, με τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κόσμο, τι επιχειρήσει, οργανώ... μη κυβερνητικέ οργανώσει και κυρίω με του Ευρωπαίου πολίτε, ε, που είναι σημαντικοί χρήση των πληροφοριών μας. Η υπηρεσία λοιπόν δραστηριοποιείται σε ένα τομέα ο οποίο ε, δεν περιορίζεται στου λαμβάνοντε αποφάσει και του πολιτικού, αλλά περιλαμβάνει και του Ευρωπαίους πολίτε, και γι' αυτό λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση στι πληροφορίε και τα έγγραφά μα. Σύμφωνα με, τα τελευταία, ε, με ένα από τα τελευταία βαρόμετρα οι πολίτε ε, επιθυμούν, να είναι, ενημερωμένοι και να συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων για θέματα τα οποία αγγίζουν την καθημερινή του ζωή. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα, η εφαρμή του κανονισμού 1049 του 2001 ε, ε, ε, διευρύνθηκε ε, και στην δική μας υπηρεσία με απόφαση τρο, αναθεώρηση του εσωτερικού του ε, συστατικού μας κανονισμού το 2003. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας υιοθέτησε το 2004 κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού 1049, τους οποίους σας υποβάλλω σε παράτημα. Το 2004 το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας μας υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Διοικητικής Συμπεριφοράς για να διασφαλίσει την διαφάνεια, την ε, αξιοπιστία και την διάβια στην λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ε, είναι ένα προϊόν αυτός ο κώδικας του Ευρωπαϊκού ε, Διαμεσολαβητή που διαχειρίζεται τις σχέσεις μας με το κοινό. Στην πράξη όλα τα έγγραφά μας είναι διαθέσιμα ε, μέσω ενός ε, ηλεκτρονικού δημόσιου μετρό με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 4 του 1049. Ε, ένας ε, νομικός είναι υπεύθυνο για την, το χειρισμό των ετοιμάτων πρόσβασης των εγγράφων και συμμετέχει πολύ τακτικά σε ε, σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνει Γενική Γραμματεία της Κομισιόν. Ε, οι επίσημες, ε, τα επίσημα αιτήματα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα ε, είναι λίγες, λίγα στην πράξη. Αφορούν περισσότερο διαδικασίες διαγωνισμών Con προμηθειών ή ε, ε, ε ανακοινώσει πρόληψη προσωπικού. Το σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση του κανονισμού 1049 σύμφωνα για την προσαρμογή του στην Συνθήκη Λισαβόνα ε, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 15.3 τη Συνθήκη Λισαβόνα, ε, είμαστε υπέρ αυτή τη επικαιροποίηση, γιατί εμεί ήδη την έχουμε εφαρμόσει από το 2003. Ε, πολύ ε, πρόσφατα μα ενημέρωσε η Κομισιόν για την τελευταία τη πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού 1049 που θα επισημοποιήσει την δυνατότητα πρόσβαση ε, στα έγγραφα τη ε, ε, υπηρεσία, ενώ ο αρχικό κανονισμό είχε προβλέψει μόνο το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Όλε οι τροποποίησει του 1049 που ε, ε, συζητώνται αυτή τη στιγμή έχουν ως στόχο την βελτίωση τη ε, διαφάνεια και ε, ε, και θα τι εφαρμόσουμε αμέσω μόλι υιοθετηθούν. Ε, επίσης ε, εφαρμόζουμε τον κανονισμό 1367-2006 όπως σας είπα αφορά την εφαρμογή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης των διατάξεων της Σύμβασης του Άρχου σε ό,τι αφορά την, προσφυγή, την ε, πρόσβαση στις πληροφορίες για το περιβάλλον και τη συμμετοχή του κοινού στην δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος. Στην πράξη αυτές οι αιτήσει, αυτά τα αιτήματα είναι πολλά και γίνονται κυρίως ε, μέσω της διεύθυνσής μας στο ίντερνετ αυτή που βλέπετε στην οθόνη. Ε, αυτό το, αυτός ο ιστότοπος ε, είναι ένας πολύ πλούσιος ιστότοπος για θέματα περιβάλλοντος. οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν εκεί πληροφορίες αλλά και μπορούν να θέσουν και ερωτήματα μέσω αυτού. Όλες οι εκθέσεις, οι συνθέσεις, συνόψεις και άρθρα ε, μπορούν να κατέβουν από το ίντερνετ ε, χωρίς ε, κανένα αντίτιμο. Αυτή θα βρείτε μάλιστα την έκθεσή μας για την πενταετή μας έκθεση, την τελευταία πενταετή έκθεση για το κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2010 ενώ κάποια άλλα πράγματα, στατιστικές να σας πω για το site μας, 300.000 επισκέψεις το μήνα, ε, είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα site μεταξύ των όλων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών το δικό μας. Ε, οι επισκέψεις προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία κατά κύριο λόγο ε, και το, περιβάλλον, το περιεχόμενο του site μας ε, είναι διαθέσιμο με την άδεια Creative Commons σε αυτή τη διεύθυνση την οποία βλέπετε. Ε, τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ε, είναι προσιλωμένη στην ε, διαφάνεια ε, που δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα που είναι απαραίτητα και χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ε, με την αναδιατύπωση του 1049 θα συνεχίσει να κάνει και ακόμα πιο διαθέσιμα τα έγγραφά της μέσω συστημάτων πιο φιλικών προς το χρήστη ε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε το κοινό και τον Ευρωπαίο πολίτη να βρει απάντηση στις καθημερινές ερωτήσεις σε θέματα περιβάλλοντος και να βοηθήσει και την εκπαίδευση του κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου για την παρέμβασή σας. Χαίρομαι που μπορώ να σας καθησυχάσω λέγοντάς ότι το Κοινοβούλιο δεν θα κινηθεί εντός να αναδιατυπώσεως. Είναι κάτι που διαβιβάστηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της πρώτερης θητείας του Κοινοβουλίου και είναι κάτι που υποστηρίζει και ο παρόν Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών Κοιτάξτε τι έχει παράγει το Κοινοβούλιο στο έγγραφο τοποθέτησής του. Είναι ένα έγγραφο με τρεις πίνακες. Μάλλον πρέπει να φορέσω και τον άλλο φακό επαφή μου. Ε, δίνει μια σαφή ιδέα της νοοτροπίας του Κοινοβουλίου. Όταν λέω το Κοινοβούλιο, αναφέρομαι στην πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Όχι, δυστυχώς, σε όλε. Σε όλου του βουλευτέ. Έχουμε ένα-δύο λεπτά για συντομότατες ερωτήσεις ή σχόλια. Η Δίετρη. ευχαριστω θα είμαι σύντομη. Να επανέλθουμε σε κάτι άλλο για την Europol. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούστηκαν. Για την Europol λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα που τίθεται. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις διαβαθισμένες πληροφορίες αλλά και τις υπηρεσίες πληροφοριών και τον έλεγχο των υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών. Ε, εγώ δεν θα υποστήριζα τον περιορισμό της προσβάσεως της Europol μόνο στα διοικητικά έγγραφα. Πρέπει να το δούμε στα πλαίσια της εταιρικής στρατηγικής, όπου υπάρχουν πολλοί φορείς που συνεργάζονται, που αποκτούν και εμπιστευτικές πληροφορίες. Είναι πολύ ευρύτερο το όλο θέμα. Κάτι άλλο. Το θέμα των εμπιστευτικών εγγράφων είναι κρισίμου σημασία. Συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας. Υπάρχει υπερβολή, υπάρχει υπερβολή στη διαβάθμιση των εγγράφων, πιστεύουμε. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβαίνει στα κάτι μελη στι ΗΠΑ. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και υπάρχει ε, τεράστιο ποσοστό υπερβολή όσον αφορά τη διαβάθμιση των εγγράφων. Ε, και είναι σαν χιονοστιβάδα. Λίγα έγγραφα ε, θεωρούνται ε, απόρριτα, άκρως απόρριτα και μετά ακολουθούν άλλα σαν χιονοστιβάδα από αυτά, που προέρχονται από αυτά. Είναι και το άλλο θέμα που αποκαλούν στις ίπα ε, η κούραση ε, ή μάλλον κόπωση που έρχεται από τον υπερβολικό έλεγχο, κάτι που διαδίδεται, διάχυση του ελέγχου από πολλούς φορείς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί στα πλαίσια της αναδιατυπώσεως του, του κανονισμού. Ευχαριστώ, Χέλεν. Εάν μπορείς να είσαι πολύ σύντομη. Σε δύο στοιχεία θα αναφερθώ. Η ανησυχία για τον ορισμό του εγγράφου, για τη διαγράφηση του εγγράφου. οι πληροφορίε που είναι σε ψηφιακή μορφή ίσω δεν είναι απαραίτητα προσβάσιμε. Συγχαίρουμε την Υπηρεσία Περιβάλλοντο για τα δημιουργικά σχόλια και την προσέγγιση αυτή που ακολουθήθηκε. Στην παρέμβασή μου αναφέρθηκα ακροθυγώ στο λογισμικό ε, που είναι ανοιχτό, open source. Ε, είναι πολύ καλό πληροφορίε που συλλέγονται από το κοινό να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ευχαριστώ, Έλεν. Δεν χρειάζεται να δοθούν άμεσα απαντήσεις σε αυτά που αναφέρθηκαν. Έχουμε 3,5 λεπτά για τα καταληκτικά σχόλια των τριών εισηγητών που είναι εδώ. Η Heidi Hautala είναι εισηγήτρια όσον αφορά την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 1049 και η Νέλη για την Εμάκη είναι συνεισηγήτρια μαζί με μένα όσον αφορά το θέμα της αναθεωρήσεως να σας γνωστοποιήσω κάτι, αν δεν το ξέρετε ήδη. Θα υπάρξει συνέντευξη τύπου, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου επί του θέματος και επί των όσων υπόθηκαν σήμα το πρωί στις 13.30 νομίζω, μία μισή, πράγματι στη συνηθισμένη αίθουσα. Και θα ήταν παράληψή μου να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τη γραμματεία και το προσωπικό του για όλη τη δουλειά που έκαναν για τη διοργάνωση αυτής της ακροάσεως και το προσωπικό της πολι των γραμματιών των πολιτικών ομάδων και τους ευρωβουλευτές, το προσωπικό των ευρωβουλευτών. Λοιπόν, σας παρακαλώ να δείξετε την εκτίμησή σας προς όλους αυτούς που ανέφερα. Λοιπόν, στο τέλος, τι, πώς μπορώ να ανακεφαλαιώσω τα σε υπόθηκαν. Να πω ότι εκείνοι που είπαν ότι η αναδιατύπωση ή η πλεον πρόσφατη πρόταση ήταν τα μόνα μέτρα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε όσον αφορά τον 1049, αν δεν είχαν παρακολουθήσει συνεδρίε Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών επί σειρά ετών, με το που ήρθαν σήμερα το πρωί και μόνο θα είδαν ότι μία απλή αναδιατύπωση ή ένα ανακάτεμα με ε, την νομοθεσία λόγω της διαστάσεως της ε, συνθήκης της Αβώνας δεν ε, αρκεί. Είναι ό,τι πειράζουν από αυτά αποτελεί προσβολή στη συμμετοχική δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά και δίνω το λόγο στην Νέλη για την Εμάκη. Ευχαριστώ, Μάικλ. Δεν νομίζω ότι έχω άλλα σοφά λόγια να προσθέσω ή να, ε, να προσθέσω τη σοφία των όσων ακούστηκαν σήμερα. Α, ας πω δύο πράγματα. Πολλά μένουν ακόμα που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην πραγματική δημοκρατία και την πραγματική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ίσως αυτό να είναι και πιο επικοδομητικό. Καλή όρεξη, αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Χάιντι, ευχαριστώ πολύ. Άξισε ε, τη διοργάνωση ε, της αυτή οι ακρόαση ακούσαν οι πολλά πράγματα που θα του τροφοδοτήσουν στι συνεχιζόμενε προσπάθειές του που ξεκίνησαν από παλιά. Ο ρόλο μου είναι να εξετάσω την εφαρμογή, την πρακτική που ακολουθείται, όπω είπε και ο Μάικλ. Ήταν πολύ πλούσια, στο ο Η εξέταση των διαφόρων περιπτώσεων, των υποθέσεων και πώ οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών ε, ζήτησαν την πρόσβαση στα έγγραφα και πώ την αρνήθηκαν επί βάσεως ε, ε, τι, ποιοι ήταν οι λόγοι για την άρνηση και πώς έφτασε η υπόθεση στα δικαστήρια στο διαμεσολαβητή. Ελπίζω α, από όσα υπόθηκαν να, να αντλήσω κάποια έμπνευση και να δω πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εφαρμογή, την εκτέλεση, την υλοποίηση του κανονισμού και αυτό σχετίζεται και με τη μορφή που θα αποκτήσει ο κανονισμός για να ταιριάζει 100% με τις συνθήκες της Λισαβόνας και το σχετικό πλαίσιο. Ξέρω τώρα καλύτερα ότι οι καθυστερήσεις όσον αφορά τις αιτήσει, τα πω αιτήσει είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, τα ακούσαν πολλούς και η πρόσβαση τρίτων μερών, το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι είναι ενοχλητικό. Επί δεκαετίες αντιμετωπίζουν το θέμα και τα κράτη-μέλη φέρονται σαν να μην αποτελούν ένα τμήμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να μην δημιουργούν μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι εξωφρενικό και το επί 15 χρόνια αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα, πρέπει να βρούμε λύση. Ποιο είναι το κατάλληλο βήμα, ίσως πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Διαμεσολαβητής. Το θέμα των εξαιρέσεων δεν καθορίζεται επακριβώς, χρειάζεται πιο ακριβής ορισμός ε, στα διάφορα βήματα προβληματισμού. Εγώ θα εξετάσω τα θέματα των διεθνών εγγράφων και με τα χαράς άκουσα τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ίσως έχουμε νέα, νέο έδαφος εδώ, νέα περιθώρια να ανοίξουμε κάπως και τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Οι νέοι οργανισμοί είναι αρκετά ανοιχτοί, ακόμα και η Frontex και πιστεύω ότι η Ζάκ Χαρίσου είναι μέλος της ομάδας εργασίας για τις ε, πληροφορίες την ενημέρωση στο Συμβούλιο και εκπροσωπούσες μια ανοιχτή φιλική χώρα. Ε, έχεις, έχεις ένα λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, το ξέρω. Πάντα το λέγαμε, Φιλανδία και Σουηδία το 1766 θέσπισαν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Είμαστε υπερήφανοι για την παράδοση και χαιρόμαστε πολλά από αυτά τα στοιχεία μεταφέρθηκαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στους ευρωπαϊκούς φορείς. Χάρηκα από αυτά, με αυτά που άκουσα από τη Frontex τη Europol και πρέπει να επανέλθουμε και στο θέμα των βάσεων δεδομένων. Εν γέννη πιστεύω ότι ο κατάλογος των εξαιρέσεων καλύπτει τις περιστάσεις που περιγράψατε. Κανεί δεν θέλει να πειράξει ε, ή να, είναι, να κινηθεί με τρόπο επιβλαβή προς επιχειρήσεις της Europol. Αλλά μας άρεσε να, ακούμε, να ακούσουμε ποια είναι η σκέψη ε, της Europol. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε συνεισηγητά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Να κλείσω κάτι από την απόφαση για την πρόσφαση πληροφορίες που αναφέρθηκε. Το Συμβούλιο έχει κάποιους καλούς εκπροσώπους. Αλλά αυτή ήταν η, η άποψη, η, γνωμοδότηση. Αν η δημοσίευση των τοποθετήσεων έχει γίνει, θα δημιουργεί το σύγχυση. Προσέθεσε, και εδώ μιλάμε για τον κόσμο του Συμβουλίου, τι είπε, προσέθεσε Πώς θα μπορούσε να είναι ειλικρινέ και ανοιχτό το Συμβούλιο αν συνεχώς φοβόταν ότι οι συζητήσεις του επί το θέμα του θα μπορούσαν να δημοσιευτούν επί συγκεκριμένου θέματος. Να λοιπόν για την ειλικρίνεια. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ που ήρθατε.